faut que je Αρχίζουμε. Καθίστε παρακαλώ. Ο κύριος Φίσα βλέπω ότι βιάζεται. Βλέπω ότι είμαστε πολύ άριθμοι, σχολιάζει η Πρόεδρος. Καλή σας μέρα λοιπόν όλοι. Αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Πριν από το σημείο 4... που είναι οι ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Η Επιτροπή θα μας ενημερώσει για τις προθέσεις της όσον αφορά την προετοιμασία τεσσάρων νέων ανακοινώσεων. Εξάλλου, το σημείο μας 6 που έχει να κάνει με το σχέδιο Συμφωνίας Σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής βγαίνει από την ημερήσια διάταξη. Η συγκεντριά μα η κυρία Γκρέσ, θα μας παρουσιάσει το θέμα τη ε, αργότερα και το νομοθετικό και το μη νομοθετικό τμήμα στην επόμενη συνεδρίασή μας. Αύριο, 19 Ιουνίου, προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κλάου Σόρενσον όσον αφορά τις σημερινές ανθρωπιστικέ κρίσει. Θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε και έναν δεύτερο μιλητή αύριο που είναι ο κύριος Ζόρζ Όκοτ Όμπο που είναι ο Διευθυντής για την Αφρική της ΥΠΑ ε, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις προοπτικές και τις δράσεις του ΟΗΕ στα πλαίσια των ε, σημερινών κρίσεων τόσο στην Αφρική ε, στην Αφρικανική Υπηρολόκληρη όσο και πιο συγκεκριμένα στο Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής αλλά και στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν. Έχετε μήπως παρατηρήσεις ή τροποποίησεις να προτείνετε. Όχι από ό,τι βλέπω. Ωραία, συνεπώς η τροποποιημένη μας ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Θα έχετε πάρει τα πρακτικά της συνεδρίασής μας της 14ης Μαΐου. Έχετε παρατηρήσεις. Αν ναι, να ενημερώσετε τη γραμματεία παρακαλώ πριν τη λήξη της συνεδρίασης αυτής. Αλλιώς τα πρακτικά εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στις συστάσεις των συντονιστών. Τις έχετε πάρει. Ε? Βασιζόμαστε λοιπόν στις αποφάσεις των συντονιστών της 24ης Μαΐου 2012. Έχετε παρατηρήσεις. Εάν ναι, ενημερώστε πάντα τη γραμματεία πριν αποτελήξει τη συνεδρίασή συνεδρίασής μας αυτής. Αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα τα αποτελέσματα αυτά. Στη συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμεί να μας παρουσιάσει τέσσερις ανακοινώσεις πάνω στις οποίες αρχίζει να δουλεύει. Πρόκειται για την ανάπτυξη και συνεργασία, έτσι. Είναι στα αγγλικά εδώ, έχω κάτι, δεν ξέρω να το διαβάσω στα αγγλικά, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ενημερώσει για τις ανακοινώσεις της αυτές. Συνεπώς, το λόγο έχει η κυρία Κατρίν Μετεβέντιγεν, έτσι. Ελπίζω να μην το σφαξα το όνομά σας. Για όσο χρόνο χρειάζεστε. Είσαστε πολύ τυχεροί, δεν είναι πάντα έτσι να ξέρετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέψτε μου να σα ενημερώσω για τέσσερα σχέδια ανακοινώσεων τα οποία εκπονούμε αυτή την εποχή υπό την ευθύνη του Επιτρόπου Πίλμπαξ. Πρώτον, έχουμε μια πρώτη ανακοίνωση για την ε, μετάβαση, κάτι το οποίο θα εγκρίνει η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012. Μια άλλη για την κοινωνική προστασία που πρόκειται να εγκριθεί τον Αύγουστο του 2012. Μια τρίτη είναι όσον αφορά την ε, επιστηστική βοήθεια που πρόκειται να εγκριθεί το Σεπτέμβριο του 2012 και έπειτα πρόκειται κάτι για, την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που πρόκειται να εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2012. Το πρώτο που έχει να κάνει για την μετάβαση για μεταρρυθμίσεις. Είναι στοιχείο κλειδί αυτό όσον αφορά την ε, σταθερότητα επιτόπου και την ευημερία του κόσμου. Άρα είναι και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν μπει σε μία διαδικασία μεταρρυθμίσεων, αλλά που χρειάζονται ε, επιπλέον δουλειά για να επιτευχθεί επιπλέον πρόοδος και έτσι μεταρρυθμίσεις να φανούν και στην πράξη. Άρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Η ανακοίνωση αυτή δηλαδή δεν αναφέρεται, δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευάλωτες χώρες ή με τις χώρες εκείνες οι οποίες ζουν κάτω από ένα καθεστώς ε, διενέξεων σειράξεων. Στόχος είναι η ανοικοδόμηση της σχέσης κράτους με τους πολίτες που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και σε μια προοπτική για το μέλλον της κάστοτε χώρας. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια νέα πολιτική με την ανακοίνωσή μας, αλλά να βελτιώσουμε την συνοχή υπέρ της δημοκρατικής μεταπολίτευσης σε τρίτες χώρες. Η ανακοίνωση θα εντοπίζει τους τομείς εκείνους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να ενισχύσουμε ε, την, ε, τις μεταρρυθμίσεις και προκειμένου αυτές να μπορέσουν να είναι πιο βιώσιμες. Βασιζόμαστε στις εμπειρίες βέβαια των ε, χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δέκα χρόνια, τις δικές τους εμπειρίες δηλαδή από μια αντίστοιχη μεταπολίτευση. Βασιζόμαστε λοιπόν και στο μέσο γυτνίασης και σε κάθε είδους πολιτική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Αυτά για την πρώτη μας ανακοίνωση, για την μεταπολίτευση. Δεύτερη ανακοίνωση που έχει να κάνει με την κοινωνική προστασία. Θα είναι έτοιμη τον Αύγουστο του 2012. Υπενθυμίζω ότι έχουμε την Agenda for Change, η οποία ζητούσε μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος αυτού με υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και κοινωνικές υπηρεσίες υπέρ μιας πιο συνολικής ανάπτυξης που να βοηθάει ώστε οι πολίτες να μπορούν να χαίρουν του πλούτου στο σύνολό τους. Η ανακοίνωσή μας λοιπόν ανταποκρίνεται σε κάποιους σημαντικούς πολιτικούς στόχους που αναφέρονται στην Agenda for Change, την Agenda για την αλλαγή δηλαδή. Πρόκειται για τις συνθήκες μιας πιο ισχυρή ανάπτυξης με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πολιτική απάντηση στις αναδυόμενες χώρες. Ε, βασιζόμαστε επίσης στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου και τη αστάθειας των τιμών, αλλά και της οικονομική κατάστασης έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Η στιγμή είναι πολύ κατάλληλη για χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στην απασχόληση ή στην πολιτική αστάθεια και που κινδυνεύει να οδηγήσει σε κοινωνίες δύο Υπάρχει η ανατμία του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίε υγεία. Αυτό θα το προσέξουμε όλο ιδιαίτερω. Θέλουμε φυσικά να είμαστε ρεαλιστέ. Κανένα δεν περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την υγεία ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Το μήνυμά μα δεν είναι διεθνέ, είναι εσωτερικό. Θα μελετήσουμε πώ οι χώρε αυτέ μπορούν να κατανείμουν καλύτερα τον πλούτο τους και πώς μπορεί να υπάρχει μια πιο στενή σχέση με, τις, ε, με τα έσοδα της ε, χώρας. Κάτι που έχει άμεση σχέση βέβαια και με τα συστήματα φορολόγησης των χωρών αυτών. Η ανακοίνωσή μας αυτή έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με το κοινό. Έχουμε πάρει 135 απαντήσεις από 8 διαφορετικές χώρες, από διάφορες διεθνείς οργανώσεις, Ηνωμένα Έθνη, ΕΝΣΕΦ, η Διεθνής Τράπεζα Εργασίας και από διάφορους εταίρους με κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και από το κοινό γενικά. Έγιναν διαβουλεύσεις επίσης και στις Βρυξέλλες με διάφορες χώρες μέλη και τέλος είχαμε και συνεδριάσεις στο εξωτερικό με αξιωματούχους από διάφορα Υπουργεία Οικονομικών, Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και με κοινωνία των πολιτών στην ε, Αφρική αλλά και στον Ειρηνικό. Ε, Καζαπλάκα, Μπαγκό κλπ. Έχουμε στη δρίτη μας ανακοίνωση για το Σεπτέμβριο του 2012. Έχει να κάνει με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η ανακοίνωση αυτή επίσης θέλει μια πιο συνολική προσέγγιση, πιο αποτελεσματική για τη συνεργασία μας με τις οργανώσεις αυτές. Ε, τονίζουμε ιδιαίτερα τι συμβαίνει στην κάθε χώρα, βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες και της κάθε χώρας αλλά και του κάθε τέρου της οργάνωση δηλαδή. Καλύπτουμε τις, κοινο... τις οργανώσεις της των πολιτών στα πλαίσια της γυτνίαση, στα πλαίσια της διεύρυνση και υπάρχει φυσικά συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση. Η ανακοίνωσή μα βασίζεται στο διαστρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις τοπικέ οργανώσει, και θα λαμβάνουμε υπόψη μα και τα συμπεράσματα τη Agenda for Change. Θα βασιστούμε επίσης στην ατζέντα για την δημοσιονομική στήριξη και γενικότερα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στη διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου. Πάω πολύ γρήγορα, λέει ο Μιλήτρια. Πήραμε 315 απαντήσεις από ολόκληρο τον κόσμο. Δέκα αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν διαβουλεύσεις με τις τοπικές οργανώσεις. Είχαμε μία διαβούλευση με περίπου 73 εκπροσώπους τοπικών οργανώσεων, τοπικών αρχών και χωρών μελών στα πλαίσια του Φόρουμ για τις Πολιτικές Ανάπτυξης που έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου. Αναλύουμε τώρα τις απαντήσεις και τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα του διαρθρωμένου διαλόγου και μας υποδεικνύουν διάφορες πρακτικές και διάφορα στοιχεία κλειδί οποία είχαμε, στα οποία είχαμε ήδη καταλήξει. Ζητάει ο κόσμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει ανευνοϊκό πλαίσιο για τις οργανώσεις αυτές, να υπάρχει μια ισχυρή πολιτική δέσμευση. Μας ζητάει επίσης να διευθρώσουμε ακόμα περισσότερο το διάλογό μας μαζί τους μέσω μιας πιο διαρθρωμένης ενημέρωσης και μας ζητάνε επίσης μια κατάλληλη χρηματοδότηση η οποία να είναι γνωστή εκ των προτέρων και μας ζητούν επίσης να βοηθήσουμε και στην κατάρτιση των οργανώσεων αυτών από την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα θέματά τους. Έρχομαι Τώρα στην τελευταία μας ανακοίνωση. Α, η προηγούμενη, όπως σας είπα, Οκτώβριο 2012 θα δημοσιευθεί και έρχομαι τώρα στην τελευταία μου ανακοίνωση. Στόχος της είναι να παρουσιάσει μια συνολική προσέγγιση αποτελεσματική, ελαστική και μακροπρόθεσμη που να βασίζεται στις ε, αλλαγές θέματα επισητιστικής βοήθειας. Τώρα, γιατί χρειάζεται μια τέτοια ε, ανακοίνωση. Το ζήτησε πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο στις 14 Μαΐου που μας πέρασε. Resilience είναι ο όρος. Τι ακριβώς εννοούμε. <clears throat> Πρόκειται για την, αντοχή. Ε, για την αντοχή. Πώς δηλαδή ένα υλικό αντιστέκεται ε, στα σοκ. Εδώ θέλουμε ακριβώς την αντίσταση μιας κοινωνίας, μιας περιοχής, μιας χώρας, έτσι ώστε εφόσον υπάρξουν παράγοντες ε, σοκ, η στρες να μπορεί να αντισταθεί. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε όλα τα φόρουμ που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Ο όρος αυτός λοιπόν αντοχή. Αντοχή όσον αφορά την επιστημική βοήθεια λοιπόν. Αυτή είναι η ανακοίνωσή μας και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στα μαθήματα που έχουμε πάρει σχετικά με την ανθρωπιστική και επισητιστική βοήθεια από την υποσαχάρη Αφρική όταν βρέθηκε σε δύσκολη επισητιστική κατάσταση είτε λόγω θεομηνιών είτε λόγω έλλειψης φυσικών πόρων είτε λόγω σειράξεων, αύξησης των τιμών των τροφίμων κλπ. κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μειώνουν κατά πολύ τις δυνατότητες των πολιτών των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις και να ανακάμψουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσέγγιση μας που είναι η αντοχή είναι ακριβώς για να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος κάθε φορά που υπάρχει μια επισητιστική κρίση. Πώς θα μειωθεί η αδυναμία του πληθυσμού και πώς θα αυξηθεί η αντοχή του λοιπόν. Θέλουμε συνεπώς να λάβουμε υπόψη μας τον παράγοντα ε, της πιθανότητας μιας επιτιστικής κρίσης και την ε, σοβαρότητα αυτής. Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε ένα μέσο πρόβλεψης επικεντρωνόμαστε σε πολύ συγκεκριμένους κινδύνους. Θέλουμε όμως επιπλέον να μπορούμε από πριν να προβλέψουμε όλους τους κινδύνους που θα κάνουν πιο ευάλωτο τον πληθυσμό σε μια περιοχή, αναλύοντας τις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν ε, τέτοια φαινόμενα επισητιστικής ε, κρίσης κλπ. Παρουσιάστηκε ήδη στα κράτη-μέλη ανακοίνωση αυτή. Ο στόχος είναι να υποβληθεί στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2012 η ανακοίνωση αυτή. Υπάρχει και μια διάσκεψη για την ε, αντοχή στο Τόκιο στο, τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Ευχαριστώ. Δεν εγκαταλείπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ο κύριος Μπιλ Νιούτον Ντάν απευθύνει μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία βρίσκεται μέσα στο φάκελο και θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Νιούτον Ντάν και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Γκριν, στην κυρία Γκριν. Πρέπει να μου βάζετε όταν είναι κυρία, διότι διαφορετικά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω αγγλικά. Ευχαριστώ τον ε, ερωτούντα για την ερώτηση. Είμαι υπεύθυνη για τη Σρι Λάνκα στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και λάβαμε την ερώτησή σας για το, τα στρατόπεδα των προσφύγων στο Ταμίλ Ναντού στην Ινδία. Ε, ήμουν τον περασμένο μήνα στην Ινδία και νομίζω ότι υπήρξε κάποια παρανόηση όσον αφορά τους όρους προσβάσεως. Για να σας εξηγήσω, δεν είχαμε προβλήματα αλλά ε, οποιαδήποτε αντιπροσωπεία της ε, ΕΚΟ που θέλει να, ε, ε, να επισκεφθεί αυτά τα στρατόπεδα πρέπει να έχει άδεια και όλα τα προγράμματα τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει από το 2002 έχουν ε, χρηματοδοτηθεί τουλάχιστον και ελεγχθεί μία φορά στον κύκλο ζωή τους, γι' αυτό και μπορούμε να συνεχίσουμε να τα χρηματοδοτούμε. Υπάρχουν βέβαια οργανώσεις οι οποίες έχουν δυσκολίες προσβάσεως και αυτό διότι ε, η ε, οργάνωση αυτή δεν έχει προσυπογράψει την ε, σύμβαση και γι' αυτό δεν μπορεί ε, να συνεργαστεί με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που είναι ε, τα στρατόπεδα αυτά. Έχουμε διαπιστώσει όμως μία σημαντική βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων λόγω της βελτιωμένης ε, βοηθείας την οποία προσφέρουν οι αρχές του Ταμίλ Ναντού και από το τέλος ε, αυτού του έτους δεν έχει χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε εμείς στον ε, προϋπολογισμό του 2012. Υπάρχουν και άλλοι δωρητές από την Αυστραλία, από τις Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν μια προσέγγιση πιο προσφυλή στην ε, ανάπτυξη η οποία είναι καλύτερη από την ανθρωπιστική βοήθεια την οποία προσφέρει το ΕΚΟ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντηση. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καθησυχαστικό αλλά δεν ήταν αυτό που μας είπα στο Νέο Δελχή διότι ε, δεν ε, μας ε, είπατε αν πήγε κάποιος εκεί γιατί στο Δελχή μας είπε ότι κανείς δεν πήγε μας είπατε ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη και την προοδό και εφόσον σταματάτε τη βοήθεια είναι ίσως καλό. Αλλά αυτό που με ανησύχησε όταν ακούσαμε την αντιπροσωπεία της ε, ΕΚΟ ή στην, ε, στο Νέο Δελχή ήταν διότι χωρίς προστασία εκεί ε, δεν θα ήταν ε, ασφαλής η επίσκεψη. Υπάρχουν εγκληματίες, ομάδες και ε, εάν τα χρήματα αυτά καταλήγουν εις τα χέρια ανθρώπων που δεν μας επιτρέπουν έχουμε πρόσβαση εις τα στρατόπεδα, τι γίνεται με τη διάσπαση του κοινοτικού χρήματος, αλλά άπαξε σταματάμε τη βοήθεια. Νομίζω ότι και η ερώτηση και η απορία είναι περιττή. Υπήρξε μία παρανόηση διότι έχουμε επισκεφτεί τις ε, τις, ε, ε, τα, ε, τους καταβλισμούς αυτούς. Έχουμε καλύψει το 10% γιατί είναι καταβλισμοί σε 1300 χιλιόμετρα οπότε έχουμε δειγματοληπτικά επισκεφθεί τους καταβλισμούς αυτούς. Βεβαίως υπήρχαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την οικειοθελή, τον οικειοθελή επαναπατρισμό των προσφύγων στη Σρι διότι οι αρχές προσπαθούν να επιβάλλουν ασφάλεια και παρακολουθούν την πρόσβαση και ή από το Νέο Δελκή από τη Σρι Λάνκα μπορέσαμε να παρακολουθούμε και ε, μας παρουσίασαν την ενημέρωση. Μάλιστα ο υπεύθυνο για το πρόγραμμα ηχό είναι αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και ίσως μπορείτε ε, να ενημερωθείτε και να γνωρίζετε γιατί δεν ε, υπήρξε επίσκεψη. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι εδώ διαφωνούμε, λέει ο κύριος Νιούτον ε, Εντάξει, αν ε, επισκεφθήκατε τους καταβλισμούς, αλλά όταν πήγαμε τον Απρίλιο δεν υπήρξε επίσκεψη. Ίσως μετά η ερώτησή μας οδήγησε σε επίσκεψη. Ο Πίτερ μόλις είχε αναλάβει τον ε, Απρίλιο τη θέση αυτή στο Νέο Δελχή και ίσως δεν ήταν ενημερωμένος αλλά οι άλλοι αντιπρόσωποι ίσως είπαν ε, εντάξει αφού ε, επισκεφθήκατε τους καταβλισμούς και από την άλλη πλευρά ε, σαμάτησε η χρηματοδότηση έκλεισε το θέμα. Είναι βασικό να γνωρίζει, λέει εκπρόσωπο της Επιτροπής, ε, της, ε, να γνωρίζουν όλοι στο ακροατήριο ότι δεν υπάρχει διάσπαση του, διασπάση του δημοσίου χρήματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε παρακολουθήσει τις αποστολές, καθυστερήσαμε την καταβολή των πόρων γιατί θέλαμε να έχουμε διασφαλίσει ότι υπήρχε σωστή αντιμετώπιση αντιμετώπιση από τους ομολόγους μας ή στους καταβλισμούς και έχουμε εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση καταλήγει στους σωστούς αποδέκτες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπήρξε παρανόηση σχετικά με αυτή την ε, ε, ανταλλαγή. Η Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να ρωτήσουμε ε, τον ε, κύριο Πίτερ γιατί, γιατί και εγώ ήμουν εκεί και γιατί μας είπε τότε ότι δεν υπήρξαν ε, επισκέψεις. Άπαξ όμως και διορθώθηκε η κατάσταση. Νομίζω ότι ίσως ήταν μία κακή ερμηνεία ή μία παρανόηση και μπορούμε να ε, εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κλείσουμε το θέμα. Και όπως είπατε, ο κύριος Νιούτον Τζον Νιούτον Τον, με συγχωρείτε. Είναι Δευτέρα και με βλέπετε λίγο ε, να έχω δυσκολίες. Ε, ε άπαξ όμως και διεκόπη η χρηματοδότηση δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχούμε. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην παρουσίαση μίας μελέτης την οποία είχαμε ζητήσει ε, στην ε, θεματική ομάδα να εξετάσει για μια συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Σαχέλ εξετάζοντας και την αναπτυξιακή πτυχή και την ασφάλεια διότι αυτές οι δύο πτυχές ε, είναι στενά συνδεδεμένες και δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα λόγω των σοβαρών πολιτικών διαταραχών και ε, των προβλημάτων ασφαλείας ε, σε υπόβαθρο λοιμού και υποαναπτύξεως Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η κατάσταση και θα σας παρουσιάσω τους τρεις παρουσιαστές της μελέτης που θα παρουσιάσουν μία σύνοψη, τον κύριο Λουί Σιμών Ναβάρο, την κυρία Αν Ελίζα Μπεθαμέλια Χάτφιλ και τον κύριο Αλεξάνδερ Ματελέρ και τους τρεις εκπροσώπους του Ινστιτούτου ευρωπαϊκών μελετών της του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελών στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, θα σας δώσω πέντε λεπτά στον καθένα και θα ξεκινήσω με τον κύριο Ναβάρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία επισκόπηση της εκθέσεώς μας για ε, μας ανετέθη πριν από μερικές εβδομάδες αυτή η μελέτη και ε, επιπλέον θα δώσω και στους ε, άλλους ομιλητές των λόγων. Στα 7 λεπτά που μου έχετε δώσει θα σας μιλήσω για την σημασία της ε, περιοχής του Σαχέλ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των δυναμικών που αλληλεπιδρούν στην περιοχή. Λοιπόν, ε, βλέπουμε ότι ο όρος Σαχέλ αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στην νότιο πλευρά της ερήμου της Σαχάρας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ορισμός Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το Σαχέλ είναι περιοριστικός και ασαφής. Η στρατηγική αυτή λοιπόν αναφέρεται στη Μαυριτανία, στο Μαλί και στο το Ήγηρα και επίσης περιλαμβάνει μέλος, μέρος του Τσάτ και του Μπουρκίνα Φάσο έπρεπε να παρουσιάσουμε μία αξιολόγηση της στρατηγικής του Σαχέλ, οπότε δεχθήκαμε ε, τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το Σαχέλ, διότι πρέπει να κατανοήσετε ότι υπάρχει ένας ευρύς γεωπολιτικός χώρος ο οποίος οριοθετείται στο Σαχέλ και αυτό σημαίνει ότι οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν τις πολιτικές και δύο άλλων περιοχών που είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βόρειο Αφρική και τη Δυτική Αφρική. Οπότε θεωρούμε ότι προσφέρει στρατηγικό βάθος εις τη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική Αφρική και γι' αυτό επηρεάζει τη σταθερότητα των γεωπολιτικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θέλω να σας πω ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή ε, σύμφωνα με τη στρατηγική του 2011 είναι οι εξής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν στενά συνδεδεμένα στοιχεία και υπάρχει μία αστάθεια του κράτους και ε, μία οικονομική υποανάπτυξη, δηλαδή έφορο έδαφος για τρομοκρατία, παράνομη μετανάστευση και ε, οργανωμένη εγκληματικότητα και αυτά τα φαινόμενα και είναι ε, σημαντικό αυτό για μας έχουν σαν στόχο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη γενικότερα. Συγχρόνως ε, το Σαχέλ έχει πολύ σημαντικούς ορυκτούς πλούτος, ουράνιο, σιδηρομετάλλευμα και παίζει μεγάλη σημασία στους, ε, στον ενεργειακό προγραμματισμό της ε, Ευρωπαϊκής Νόσου σχετικά με την ηλιακή ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι οικονομικές και οι πολιτικές δομές για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε των απειλών που διαμορφώνονται στην περιοχή και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται. Και αυτό έχει τονιστεί επανειλημμένος στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το Σαχέλ για να συντονίσει κανείς τις προσπάθειες ασφαλείας και αναπτύξεως. Όπως όμως είπαμε στην έκθεση, ο ε, συγχρονισμός των προσπαθειών ε, είναι μεγάλη πρόκληση και το πιο βασικό θέμα που μας απασχολεί είναι ότι υπάρχει κι άλλο ένα εμπόδιο στην σταθερότητα της περιοχής και στα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή ε, και ε, μπορούμε να διαδραματίσουμε στα πλαίσια αυτά ένα πιο σημαντικό ρόλο από πλευράς στρατιωτικής βοηθείας γνωρίζοντας καλύτερα την περιοχή. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό διότι εάν δεν τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η δραστηριο... αναπτυξιακή δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή απλούστατα ε, θα ε, διαιωνίζει την ε, τα χαρακτηριστικά τα οποία οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και στην αστάθεια η οποία υπάρχει. Προτού όμως δώσω το λόγο στην κυρία Μέλια Χάτφιλτ, στη συνάδελφό μου, θέλω να σας περιγράψω βασικά τους βασικούς συμμετέχοντες σε αυτό το πλαίσιο και καταρχήν να σας πω ότι οι εξωτερικοί παίκτες εκτός δηλαδή από τον πυρήνα του Σαχέλ όπως τον καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση που παίζουν ρόλο εδώ είναι η Λιβύη και η Αλγερία και οι δύο χώρες αυτές ε, βρίσκονται από τη μία πλευρά προς την ε, Βόρειο Αφρική και από την άλλη προς το Σαχέλ. Είναι δηλαδή άμεση γείτονες της Ευρώπης ε, στο ε, το καθεστώς του Καντάφη είχε επέμβει κατευθείαν τα τελευταία χρόνια στην Μαυριτανία, στο Τσάντ, στο Μαλί, ε, μέσω των ομάδων του Αρέγ και άλλων ε, μεσαζόντων και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η Λιβύη για την περιοχή αυτή. Η Αλγερία θεωρεί ότι είναι ο φυσικός ηγέτης του Μαγκρέμ και θεωρεί ότι η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέτουν σε κίνδυνο την ε, ηγετική της θέση για την περιοχή και πιστεύουν ότι στις επόμενες ε, δεκαετίες θα εξελιχθεί η κατάσταση και μπορούμε να το συζητήσουμε πιο λεπτομερώς στη συνέχεια. Ήδη αναφέρθηκα στο ρόλο των Ηνωμένων πολιτιών που ήταν πολύ σημαντικό στα τελευταία δέκα χρόνια ιδίως στο θέμα της τρομοκρατίας διότι υπάρχει στενή σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αλγερία για την τρομοκρατία και θέλω να αναφερθώ και στην ε, ε, στο θέμα της εξορρυκτικής βιομηχανίας και της, ε, των θρησκευτικών ε, αιρέσεων που είναι ε, πολύ ριζικές εκφράσεις του Ισλαμισμού. Πριν όμως τελειώσω σε επιτροχάδιν θέλω να αναφερθώ ποιος είναι ο σημαντικός ρόλος των ε, ε, παικτών που δεν είναι κράτη η Τουαρέγ, η Μπόκο Χαράμ, το μέτωπο Πολυσάριο ε, και τη σημασία των δικτύων διακινήσεως ναρκωτικών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ, Λουίς. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ περίεργη, δύσκολη η έκθεση αυτή την οποία πρέπει να συνδέξουμε, διότι το interface ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια και σας ε, εξηγήσαμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε σε μια από τις πιο προβληματικές ε, περιοχές του κόσμου Άρα τα θέματα ασφάλειας ε, έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ασφάλειας στην Λιβύη μετά τον πόλεμο, στο Μαλί, γιατί υπήρξε και ένα ε, πραξικόπημα, κάτι που δεν μας βοήθησε με την επανάσταση των του Αρέγκ στην Πουρκίνα Φάσο. Ε, το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει οι υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα φτώχειας, ε, προβλήματα στη γεωργία, προβλήματα έλλειψης ε, τροφίμων. Η ανάπτυξη αφορά επομένως Λοιπόν, προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά και εμφανίζονται και στο κείμενο που αφορά την στρατηγική του Σαχέλα η έκθεση αναφέρεται κάποιες, σε κάποιες στρατηγικές δράσεις, δηλαδή θέλουμε να θίξουμε τι πρέπει να αλλάξει τα... και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι πρέπει να αλλάξει, αλλά και πώς θα αλλάξει αυτό. Άρα το πρόβλημα δεν είναι να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξει αλλαγή, αλλά το πρόβλημα είναι πλέον και πρακτικό. Επίσης θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει αυτή τη στιγμή στη σχέση της ε, με το Σαχέλ. Και αυτή είναι η πρώτη δέσμευση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σαχέλ. Και δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ αργές γιατί μιλάμε για τις πιο φτωχές, για, την πιο φτωχ... για τις πιο φτωχές και τις λιγότερο ασφαλείς χώρες του πλανήτη μας και προσπαθούν όλες αυτές οι χώρες να ε, πετύχουν τους στόχους ε, της χιλιετίας, ε, αλλά κάθε μία από αυτές έχει το 50% του πληθυσμού της να ζει με ένα δολάριο την ημέρα και να έχει να αντιμετωπίσει και ένα πολύ κακό κλίμα γενικότερα, πολύ δύσκολη πρόσβαση στο νερό, ε, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν κρατικές πολιτικές, ε, δεν υπάρχει καμία πολιτική ισότητα μεταξύ στα δύο φύλλα, δεν υπάρχει ισότητα τα κτλ. Επομένως, το πρόβλημα είναι ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από πληθυντική μας πλευράς και η έκθεση είναι σαφής μεν, αλλά εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνει μια ε, προσπάθεια να ενισχύσουμε την ανάπτυξη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φτώχειας. Η φτώχεια είναι ενδυμική στην περιοχή, ε, υπάρχουν προβλήματα στη γεωργία, υπάρχουν προβλήματα στις αποδόσεις ε, των καλλιεργειών Επομένως πρέπει να υπάρχουν προγράμματα δράσης για κάθε μία από τις χώρες του Σαχέλ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της διατροφικής ασφάλειας. Εάν δεν υπάρχει μία πολιτική επιβίωση σε αυτόν τον χωρό, δεν πρόκειται να ε, κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί από τη στιγμή που θα εξασφαλίσουμε κάποια κάποιο ποσοστό, κάποια πιθανότητα επιβίωσης των πολιτών αυτών των χωρών, μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα και να ε, ενισχύσουμε τις κρατικές υποδομές, ε, την επαιδεία, ε, την, απασχόληση, την πολιτική ενέργεια ενδεχόμενα. Αυτό σε μια, σε μια δεύτερη φάση. Επίσης η περιφερειακή ολοκλήρωση που είναι ένα στοιχείο το οποίο επαναλαμβάνεται και στην έκθεση την EAS και στην έκθεση, εάν την έχετε διαβάσει, στην σελίδα 2021, ε, θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Το ένα είναι το φαγητό, η φυσική πόρη, γιατί μιλάμε για μια περιοχή όπου έχει εγγενώς πολύ κακές κλιματολογικές συνθήκες και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως καμία κοινωνική ή γεωργική υποστήριξη ε, για τις ε, οικογένειες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, δυσμενείς συνθήκες, ε, τις κλιματικές συνθήκες και αυτό τι σημαίνει, ότι το τελευταίο εξάμεινο ή τον τελευταίο χρόνο είχαμε 12 εκατομμύρια άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν στην περιοχή σοβαρότατους κινδύνους κακής διατροφής, για να μην πω και πείνας. Οι κλιματικές συνθήκες έχουν ε, δυσκολέψει την κατάσταση στην περιοχή. Από τη μια πλευρά έχουμε πολλές βροχές, από την άλλη έχουμε ξηρασία. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η γεωργία δεν μπορεί να αποδώσει, έχουμε πάρα πολύ μικρές αποδόσεις. Δεν υπάρχουν εισοδήματα ε, για τους γεωργούς δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης ε, το οποίο να εξασφαλίζει αυτή την περίφημη αντοχή. Τώρα, υπάρχει και, το τομέα, και ο τομέας της ενέργειας που θα μπορούσε να βοηθήσει, που θα μπορούσαμε να τον εκμεταλλευτούμε. Γιατί υπάρχουν ε, διάφορες, διάφοροι φυσικοί πόροι στην περιοχή δεν έχουμε να κάνουμε τόσο πολύ, δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα ορυκτά καύσιμα, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι, μόνο όχι βιομάζα, αλλά φωτοβολταϊκά, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή την ηλιακή ενέργεια. Ε, επίσης υπάρχουν και άλλα προϊόντα ή άλλα project που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, παραδείγματος χάρη ο αγωγό ε, ε, διάσκηση της Σαχάρα. Επίση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε μια πράσινη ανάπτυξη των χωρών της ε, Σαχάρας. Και τώρα δίνω το λόγο στον συναδελφό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αμίλια. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Οι συνάδελφοί σας παρουσίασαν την γεωπολιμική δυναμική που αντιμετωπίζει το Σαχέλ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή όσον αφορά την ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω λιγάκι σε ένα άλλο θέμα. Πώς δηλαδή αξιολογούμε την στρατηγική για το Σαχέλ έτσι όπως αυτή υιοθετήθηκε το 2011. Βάσει λοιπόν της έρευνας που έχουμε κάνει εμείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόοδος αλλά παραμένουν πολλές προκλήσεις. Βέβαια συνεχίζουμε να περιγράφουμε έτσι την επιδείνωση σε διάφορα καυτά σημεία του πλανήτη. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρόσφατα ασχολήθηκε με το θέμα. Μπορείτε να διαβάσετε διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει είτε τώρα ξεκινάνε, μπαίνουν στο αυλάκι. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω κάποια επικριτικά σχόλια εγώ για τις δραστηριότητες αυτές που ξεκινούν. Παρά τις όποιες δράσεις, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός. Εξακολουθεί να υπάρχει κατακαιρματισμός παρόλο που προσπαθήσαμε να τον αποφύγουμε. Δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε μεταξύ θεσμικών οργάνων, θα έλεγα εγώ, για το πώς πανώνται τα διάφορα κονδύλια. Είτε πρόκειται για την ανθρωπιστική κοινότητα, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε πρόκειται για εξωτερικούς, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή παράγοντες, ένα είναι το συμπέρασμα, ότι δεν ξέρουμε αυτά τα αναπτυξιακά κονδύλια πώς ακριβώς πανώνται. Δεύτερον, όπως είπε και η Αμέλεια πριν από λίγο, η επισητιστική βοήθεια μόνο μερικώς αναγνωρίζεται ως ένα στοιχείο κλειδί. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να υπογραμμίσω ότι όταν πρόκειται για επίγουσα βοήθεια, αυτή η επίγουσα βοήθεια δεν μπορεί έτσι καλώ να αντικαταστήσει τις μακροχρόνιες και μακροπρόθεσμε αναπτυξιακέ προσπάθειε. Τρίτον, και εξίσου σημαντικό, είναι το θέμα τη ταχύτητα τη εφαρμογή. Όταν το θέμα μπήκε για πρώτη φορά στην Εμερήσια διάταξη, αυτό που θέλαμε να κάνουμε η, Ευρική, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχει αποτελέσματα και τελικά ε, προληπτικά. Τελικά όμως αντί να προλάβει κάτι η κατάσταση εκεί επιδεινώθηκε. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι όσον αφορά τα κονδύλια, η αναπτυξιακή ατζέντα συνεχίζει να κυριαρχεί το πρόγραμμα δράσης στο Σαχέλ. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ θα ήθελα να πάμε λιγάκι πιο μακριά και να σκεφτούμε λιγάκι τι, πώς μπορεί να δει τις επιλογές της πολιτικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Έτσι, ποια είναι η δράση του SDP. Υπάρχει μια κρίση ασφάλειας στην περιοχή, αναμφίβολα. Είτε απορρέει από τις εξελίξεις στην Λιβύη, είτε από άλλα στοιχεία τα οποία έχουν κυριαρχήσει στην περιοχή για δεκαετίες. Έπειτα έχουμε και το, πραξικό, το πραξικόπημα στο Μαλί και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το είδαμε να έρχεται. Ήταν γνωστό δύο χρόνια. Υπάρχει και μια αποστολή ε, οικοδόμησης ικανοτήτων για τον Ήγηρα. Τώρα είμαστε στο επιχειρησιακό στάδιο Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υπογραμμίσουμε ότι οι μικρές και μη στρατιωτικές αποστολές δεν φτάνουν για να έχουμε αποτελέσματα, για να αλλάξει δηλαδή αυτό το σπιράλ που επιδεινώνει καθημερινά την κατάσταση στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές συντονισμό στρατιωτικής, για παράδειγμα, δράσης υπό την αιγίδα της Ευρώπης. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι χώρες μέλη έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιούνται στρατιωτικά. Θα ήταν προτιμότερο να υπήρχε συντονισμός υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να εξοδεύονται όλα τα αναπτυξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αποτέλεσμα και οι στρατιωτικές δράσεις να γίνονται χωριστά από την κάθε χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προβάλλει περισσότερο την δράση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι και η ταχύτητα. Ο πρωθυπουργός του Νίκερ ήταν εδώ στι Βρυξέλλε και τι είπε, είπε ότι η χώρα μου καταραίει. Και ποιο είναι το μήνυμα που μου δίνει η Βρυξέλλε, Ε, θα στείλουμε κάποιου τον Αύγουστο. Ωραία, εγώ τώρα τι κάνω όμω. Ας δούμε τώρα την περιφερειακή συνεργασία. Σε ένα βαθμό υπάρχουν διαφορετικά πλαίσια που είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Υπάρχουν δράσεις υπό τους Ευρωπαίους και υπάρχουν και δράσεις υπό τους Αλγερινούς. Εμείς υπογραμμίζουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν πολυμερείς πρωτοβουλίες και δράσεις. Και αυτό μέσω ενό δικτύου σχέσεων το Βόρειο Μαλί είναι ο πυρήνας του προβλήματος, αλλά και της λύσης. Από τις πλευράς των Αλγερινών τα πράγματα βέβαια φαίνονται διαφορετικά. Εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι μετά την εξαφάνιση του καθεστώτος του Καντάφη η Λιβύη αποτελεί σίγουρα έναν πάρα πολύ σημαντικό εταίρο και για να καταπολεμηθούν και τρομακριτικές ε, ε, δραστηριότητες, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πάντα εμπιστοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν δύο πλαίσια συνεργασίας που θα μπορούσαν ε, μεταξύ τους να κάνουν πολλά, αρκεί να μιλήσουν μεταξύ τους. Τώρα, φτάνω στα συμπεράσματά μου. Πιστεύουμε ότι διαφορετικά πολιτικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Αλγερία αποτελεί έναν απαραίτητο παράγοντα για την λύση. Και όπως είπε και η Αμέλεια πριν, υπάρχουν τα διάφορα αναπτυξιακά πλαίσια, τα οποία πρέπει μεταξύ τους να συντονιστούν καλύτερα είτε πρόκειται για προγράμματα χωρών μερών για το Σαχέλ, είτε για οτιδήποτε άλλο. Η επισητιστική βοήθεια και η πράσινη ανάπτυξη για μας πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, να είναι προτεραιότητα. Χρειάζονται επίσης δράσεις και στρατιωτικές και μη στρατιωτικές. Και πιστεύουμε ότι το πρόβλημα που τίθεται για το θέμα του προσωπικού ότι δεν αρκεί κτλ. είναι βέβαια αντιπαραγωγικό και πρέπει να λυθεί. Είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Θα περάσουμε στι ερωτήσει. Παρακαλώ, Κύριο Γκέρεν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου ζήτησε καταρχήν να γίνει η μελέτη αυτή, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντάκτες της μελέτης αυτά που μας είπαν βοηθούν να αρχίσει η συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί βέβαια πέρα από το έγγραφο το οποίο μας υποβλήθηκε. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά εισαγωγικά. Εδώ η αίθουσα είναι περίπου άδεια. Μην ξεχνάμε ότι το Σαχέλ είναι πάρα πολύ σημαντική περιοχή και είναι λυπηρό που είμαστε μόνο τέσσερις ευρωβουλευτές εδώ. Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό για μένα. Αυτή ήταν μια παρένθεση που έκανα, την κλείνω. Για να μπω στην ουσία του θέματος. Το Σαχέλ. Πηγή προβλημάτων, ασφάλεια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλιματικές αλλαγές. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία εγώ βέβαια μπορεί να μην διάβασα σε βάθος τη μελέτη σας, αλλά πάντως από αυτά που άκουσα δεν αναφέρατε στη δυναμική των αλλαγών ένα στοιχείο που πιστεύω ότι είναι πολύ ειδικό στην περιοχή αυτή. Και αυτό είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η ιστορικό ρεκόρ. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο δυναμικό δημογραφικό. Πουθενά, σε καμία περιοχή του κόσμου. Και ποτέ ανά τους αιώνες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπογραμμιστεί. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη στο Σαχέλ, να ξέρουμε ότι η ανάπτυξη ξεκινάει α, μετά το 3%. Γιατί το πρώτο 3% απορροφάται από την αύξηση του πληθυσμού. Σε εμά είναι 0,2% αυτό το όριο, ενώ εκεί είναι το 3%. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι επίσης μια περιοχή που επηρεάζεται από την Αλγερία, το Μαρόκο, τη Λιβύη, τα είπατε κι εσείς. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν ε, την κατάσταση. Και είναι και μια περιοχή στην οποία ορμάει ο καθένας που κοιτάζει τα συμφέροντά του. Κίνα για παράδειγμα ε, και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μια πολιτική που δεν είναι πάντα τόσο ευγενή όσο αναφέρεται στα έγγραφα της Κομισιόν. Δεν λέω ότι φταίει η Κομισιόν. Το θέμα είναι λοιπόν μήπως θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα κομμάτι της λύσης αντί να είμαστε κομμάτι του προβλήματος. Η Επιτροπή είναι ο μόνος μεγάλος παίχτης, ο κύριος δωρητής βασικά, όσον αφορά λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ας δούμε το έγγραφο Responsibility του Protect. Η κύρια αιτία των προβλημάτων εκεί είναι η ακραία φτώχεια, η οποία προκαλεί ανασφάλεια, αστάθεια, πηγές όλων των διανέξεων και των σειράξεων που έχουμε εκεί. Από αυτή την άποψη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν πιο συγκεκριμένα αλλά και το Αναπτυξιακό Ταμείο που διαχειρίζεται η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Στο δυναμικό αυτό των αλλαγών υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο αναφερθήκατε και το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η περιοχή αυτή να είναι ένας ιδανικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία αποτελεί ένα εργοτάξιο θεσμικών ε, αλλαγών. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες, τι βλέπει, βλέπει ότι αλλού στον κόσμο, εκεί για παράδειγμα, προσπαθούμε να πετύχουμε την ανάπτυξη αντιγράφοντας το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσατε να είχατε πει, θα μπορούσε να είναι πιο συνεκτική και να έχει ακούσει πιο προσεκτικά τον Επίτροπο τον Αρμόδιο για την Ανάπτυξη από ότι ο Επίτροπος υπεύθυνο για το εμπόριο. Υπάρχουν δηλαδή κάποια διαβήματα που γίνονται από τη δικιά μας την πλευρά που δεν έχουν συνοχή. Εγώ θυμάμαι, το 2004 ήταν νομίζω, τότε ο Μισελ είχε αναλάβει τα καθήκοντά του Επίτροπος Αρμόδιος για την Ανάπτυξη και είχε επιμείνει τότε και είχε πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν συμφωνίες οικονομικής οικονομικής-ετερικής σχέσης, έτσι τις ονομάζαμε τότε, περιφερειακού χαρακτήρα, και να αποτελέσει ο μηχανισμός αυτός ένα στοιχείο ανάπτυξης. Ενώ ο αρμόδιος για το εμπόριο επίτροπος ξεκίνησε από μια διαφορετική βάση. Έλεγε ότι η περιοχή αυτή πρέπει να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία. Μα πρέπει κανείς να αντιλαμβάνεται ότι μια διαδικασία πρέπει να γίνεται σταδιακά. Πρώτα να ενισχύσουμε σε περιφερειακό επίπεδο το εμπόριο, στα πλαίσια της ε, Οικονομικής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια της Ένωσης για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, πριν διακινδυνεύσουμε ένα πιο σημαντικό άνοιγμα στην παγκόσμια οικονομία. η οποία στην περίπτωση που εκτεθεί έτσι απότομα η περιοχή ε, κινδυνεύει να την κάνει να πληρώσει πολύ ακριβά το εγχείρημα αυτό. Είναι χρήσιμο λοιπόν να δούμε και νέες ευκαιρίες που υπάρχουν τώρα και που δεν υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Για παράδειγμα το ψηφιακό χάσμα, πώς θα καλυφθεί. Υπάρχουν προγράμματα, σχέδια που προσπαθούν να βρούνε μια λύση επειδή δεν υπάρχει υποδομή η χερσαία. Μέσω δορυφόρου. Να, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δημιουργηθούν ε, τερικέ σχέσεις δημοσίου. Εντάξει, είμαι πολιτικός και σαν πολιτικός μιλάω, έτσι, γιατί μένα δεν μου φτάνουν οι διαπιστώσεις. Ο δικός σας ο ρόλος δεν είναι να δώσετε πολιτικές συμβουλές. Εγώ όμως παρόλα αυτά θα ήθελα να σας ακούσω να, να πτήσετε περισσότερο το εξή. Έχουμε λάβει υπόψη μας αρκετά τη δυναμική αλλαγών, τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα. Και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μέσα στη διάθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει τον κατεξοχή εταίρο της περιοχής αυτή σήμερα. Μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη ταλέντα, είναι γεμάτη πλούτο. Νομίζετε ότι αν επιμένατε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση θα προδίδατε την εντολή που σας έχει δοθεί, αντί να μιλάτε περισσότερο για την κρίση η οποία πλήττει την περιοχή. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε κανείς να ξεπεράσει τις διαπιστώσεις, να πάει πιο πέρα. Και να τονίσει πέρα από τις όποιες επικρίσεις που φυσικά και πρέπει να γίνονται. Πρέπει να επικρίνει κανείς την πολιτική. Εννοείται ότι όποιος δεν κάνει τίποτα, ε, τι κριτική να του αποδοθεί. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει, έχει το κλειδί για να βοηθήσει την περιοχή του Σαχέλ. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο τον έχει η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Καταρχήν, να σας συγχαρώ κι εγώ για την έκθεση. Η, η πρώτη ερώτηση αφορά αυτά τα πολύ σωστά που μας είπατε ότι στην περιοχή υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη δημοκρατίας, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει η απόλυτη φτώχεια, υπάρχει ανεπάρκεια στην εκπαίδευση και η ευρωπαϊκή βοήθεια που πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκέρενς μπορεί να μην είναι και τόσο αθώα όπως πραγματικά μπορεί να συμβαίνει με την κινέζικη βοήθεια εξυκνίδες στην επισητιστική, στην πράσινη ανάπτυξη, στην στρατιωτική δράση, στην καταστολή, στη μη στρατιωτική δράση. Ε, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής παιδείας και της δημοκρατικής εκπαίδευσης αυτών των πληθυσμών. Σε όλα τα φόρα, σε όλα τα συνέδρια, σε όλες τις συνεδριάσεις λέγεται ότι αν δεν εκπαιδευτούν οι πολίτες προς κάποια συγκεκριμένη μορφή παιδείας, κανένα μα κανένα από όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα που λέμε δεν πρόκειται να πετύχει. Θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα του Arab Spring, όπου κέρδισαν μεν την ελευθερία τους από δικτατορικά καθεστώτα, αλλά δεν ξέρουν πώς να την διαχειριστούν αυτή την ελευθερία, γιατί δεν έχουν δημοκρατική παιδεία. Δεν το γενικεύω αυτό το θέμα, υπάρχουν και οι άνθρωποι με σωστή. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι για μένα ένα βασικό στοιχείο της ανάπτυξης μιας περιοχής. Υπάρχει καμιά προσπάθεια για την εκπαίδευση ε, των, πληθυσμών, των νέων, των πολιτών, των κοριτσιών. Γιατί λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά εκπαίδευση αν δεν εκπαιδευτούν οι, τα κορίτσια. Και το δεύτερο, μπορεί να μου λείπει κάποια μορφή πληροφόρησης, αλλά έχετε παρουσιάσει μια λίστα όπου κάποια κινήματα τα οποία εγώ γνώρισα ως απελευθερωτικά κινήματα στο παρελθόν, όπως είναι το κίνημα Πολυσάριο, ε, και κάποια άλλα ανάλογα. Δεν ξέρω πώς έχουν εξελιχθεί αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάποια φάση ήταν απελευθερωτικά κινήματα που αγωνίζονται για την απελευθέρωση της, των περιοχών. Τα έχετε βάλει στην ίδια λίστα με drug trafficking ε, networks. Ε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι και πολύ σωστό, γιατί κάπου μπλέκουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά. Το λόγο έχει ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ πολύ για τις εκθέσεις σας είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι, διότι εγώ είμαι στην Επιτροπή ΚΡΙΜ που, ε, και που εξετάζει το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή με ενδιαφέρει το οργανωμένο έγκλημα στο Σαχέλ. Μπορεί κάποιος να το καταπολεμήσει, διότι δεν υπάρχει μία τοπική οργάνωση. Ε, φαντάζομαι ότι είναι αρνητική απάντησή σας, αλλά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Και επίσης όσον αφορά το τελευταίο σημείο ήταν το θέμα της ελήψεως συντονισμού μεταξύ των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατικών προσπαθειών, διότι ποτέ δεν ακούμε ποια κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει. Ποιος δεν συνεργάζεται, ποιος παρίσταται επί Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν απαντήσω όμως ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σον Ντόιλ εν ονόματι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε, είμαι ο υπεύθυνο για την Δυτική ε, Αφρική και λυπούμε που δεν μπόρεσαν να έρθουν οι συνάδελφοί μου εδώ σήμερα αλλά η έκθεση κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετική, είναι πολύ καλά παρουσιασμένη, είναι μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση του περίπλου χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Σαχέλ και υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία υπολείπονται ε, αλλά είναι θέματα νομικά δηλαδή η, η ε, πόροι στρατιωτικοί δεν είναι κάτι που ελέγχει η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως. Μπορεί να μιλάμε για έλλειψη συντονισμού, αλλά τυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και ε, από την άλλη πλευρά κάτι το οποίο ε, ίσως δεν εμφανίζεται είναι ότι το καθεστώς στο Μαλί ε, θεωρείται ότι ήταν αποτελεσματικό και οι εκλογές που επρόκειτο να γίνουν μετά το πραξικόπημα της 20-21 Μαρτίου ε, πρόκειτο να παρουσιάσουν μια νέα ανανεωμένη και ενισχυμένη προεδρία. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή χρησιμοποίησε ε, ο στρατός για να παραλύσει ε, το, τις δυνάμεις στο Νότο και ήταν η χειρότερη ενέργεια στη χειρότερη στιγμή. Το γεγονός ότι στη συνέχεια διατηρήθηκε η παράλυση στον Παμάκο με δύο-τρεις εξάρσεις το τελευταίο καιρό και μεγάλη αμφισημία στο θέμα της ΕΚΟΒΑΣ και πολλές αμφισημίες στο θέμα των δράσεων του Μπαμάκο και ατυχώς το χειρότερο ήταν ένα αντιπραξικόπημα της προεδρικής φρουράς που ενίσχυσε τους πραξικόπηματίες και την προσωρινή προεδρία σε was να επέμβουν και να μπορέσουν να δράσουν στο Νότο. Το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας ήταν κάτι που είναι, ήταν γνωστό και στους πρώτους μήνες του έτους έπρεπε να δούμε πώς θα το οι προσπάθειες και ένας από, τους, από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν σήμερα ήταν ακριβώς να συζητήσουμε με τους ηγέτες της περιοχής να δούμε πόσο θα πρέπει να υπάρξει ε, κάποια ε, επιχείρηση και ε, η σημασία της ε, επιστημιστικής ασφαλείας είναι πολύ πιο σημαντική και ένα μέρος του προγράμματος θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις από όταν καταρτίστηκε αυτή η έκθεση τον Απρίλιο, είναι ότι καταρχήν η σημασία της Αλγερίας αναγνωρίστηκε από τα κράτη-μέλη, συζητήθηκε σε διάφορες συζητήσεις όπως π.χ. την περασμένη εβδομάδα και δεν είναι απλώς μία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών και των βασικών άλλων παικτών ότι η ΕΚΟΒΑΣ δεν ήταν πολύ αποτελεσματική ε, σαν ε, μεσάζων αλλά υπήρξε και κάποια κινητοποίηση η οποία κατέληξε ε, σε μία σύγκρουση στη συνάντηση του Αμπιτζάν μεταξύ των Αφρικανών συμμετεχόντων του του PSC και ε, όπου είχαν καταρτιστεί ορισμένες αρχές γύρω από την ΕΚΟΒΑΣ ε, ε, με την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ για να υπάρχει μεγαλύτερο κύρος στις αποφάσεις που λαμβάνονται και να αντικτατροπρίζεται η προσπάθεια να απευθυνθεί κανείς στον ΟΗΕ ώστε η ΕΚΟΒΑΣ να μπορέσει να προβεί σε μία κίνηση ε, ένοπλη εάν ε, είναι δυνατόν και χρειαστεί. Ε, παρόλο που λέμε υπόρους διότι στο βορρά ε, χρειάζεται μία ενίσχυση η οποία δεν υπάρχει θα πρέπει να υπάρχει στήριξη της εξωτερικής ε, των εξωτερικών συνεργατών που δεν έχουν εκδηλωθεί αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι προσπαθίζουμε, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα διότι η ΕΚΟΒΑΣ πρέπει να δει τι είναι εφικτό και να δημιουργήσουμε μία αξιόπιστη δυνατότητα αντιμετωπίσεως της κρίσεως κατά τρόπον ώστε να μπορέσει κανείς να ενισχύσει αυτούς που αντιμετωπίζουν τους ταραξίσεις στο βόρειο φορά. Ε, Υπήρξε μια συν, συνάντηση στις 7 Ιουνίου και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Βορρά να μην γίνουν διαπραγματεύσεις με, κάποιον ο οποίος δεν δέχεται ε, την ακαιρεότητα του Μαλή στο σύνολό του και να μην υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες. Επιπλέον η ΕΚΟΒΑΣ, η Αφρικανική Ένωση και άλλοι συνεφώνησαν για ακυρώσεις ιδίως ε, οικονομικές οι οποίες ε, είχαν αποτέλεσμα στην αρχή άμεσα μετά το πραξικόπημα και θα έπρεπε κανένας να πείσει τον προηγούμενο πρόεδρο τον Τζουκούμ Ταρέ να επιστρέψει από το Παρίσι και να ξεκινήσει και πάλι προσπάθειες αλλά όλες ε, οι προσπάθειες έχουν αποτύχει λόγω της ελλείψεως τοπικής ηγεσία, το οποίο είναι ένα σημείο που προσπαθούμε να επιλύσουμε σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ, θα ξαναδώσω το λόγο στους συντάξαντες τη μελέτη για να μπορέσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν προσπαθώντας να σας πείσω να είσαστε σύντομοι ενώ μέτρο του δυνατού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις σε θέματα τα οποία ετέθησαν και ορισμένα ίσως θα πρέπει να εξεταστούν πιο λεπτομερώς από τους συναδέλφους. Νομίζω κύριε Γκέρενς ότι πολύ σωστά ε, τονίσατε τη σημασία της ε, δημογραφικής αναπτύξεως της περιοχής που ισχύει όχι μόνο για το Σαχέλ αλλά για όλη τη Δυτική Αφρική και είναι θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι αυξάνεται ο πληθυσμός, αλλά αυτό σημαίνει ότι το, η έκθεση δεν το τονίζει αρκετά. Πιστεύω ότι αυτό δεν καταρρύπτει τη λογική της εκθέσεως, αλλά η γρήγορη δημογραφική ανάπτυξη είναι και απειλή και ένας αυξητικός παράγων για την περιοχή για να αυξήσει τη φτώχεια, την αστάθεια, τις παράνομες μετακινήσεις πληθυσμών αν ε, δεν καταφέρουμε εκ των έξω να ρυθμίσουμε τα πολιτικά θέματα θέματα. Αλλά ε, η ευημερία, εάν επιτευχθεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, που θα στηρίξει την ε, ανάπτυξη, εφόσον εμείς έχουμε δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη, πρέπει να ισοσκελίσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την πληθυσμιακή ανάπτυξη στην οποία περίπτωση αν ισοσκελιστούν αυτά τα δύο θα μπορέσει να είναι πολύ επιτυχές το εγχείρημα. Ε, όσον αφορά το πολυσάριο, το πολυσάριο είναι, έχει περιληφθεί στους μη κρατικούς παράγοντες και είναι ενεργό στην περιοχή. Εγώ αναφέρθηκα στο Πολυσάριο σαν κοινωνικό ε, φαινόμενο, όχι τρομοκρατικό, παρόλο που υπάρχει αλληλεπίδραση με την ομάδα που διακινεί τα ναρκωτικά. Δεν θεωρούμε ότι είναι απλώς ένα ε, κοινωνικό, πολιτικό ε, κίνημα και απελευθερωτικό Όπω όπως λέμε στη σελίδα 16 και θα περιοριστώ σε αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, χωρίς μικρόφωνο. το κάνω αυτό. Μιλάμε και για τα άλλα κινήματα που έχουν να κάνουν ε, με την παράνομη διακίνηση. Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση. Ναι. Αναφέρεται σαν μη κρατικό φορέα, γι' αυτό. Το σχόλιο εκτό μικροφώνου. Είναι θέμα κατηγοριοποίησης, αν θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που δείχνουν ακριβώς και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι βουλευτές γιατί είναι όντως και πολύ ενδιαφέρουσα και η περιοχή. Θα κάνω μια σύνοψη και θα απαντήσω και στις ερωτήσεις που μου φάνηκαν όλες ενδιαφέρουσες. Τώρα, κατά πόσον η Κομισιό είναι ένας βασικός παίκτη, αν θέλετε, όντως η υπηρεσία της Κομισιό είναι ο φορέας παρέμβασης στο Σαχέλ και όπως είπατε και εσείς ο στόχος, ο βασικός μας στόχος είναι ο περιορισμός της φτώχειας. Αυτό είναι και ένα στοιχείο σταθεροποίησης. Δεν χρειάζεται να, πούμε και να βρούμε πολλά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε τον στόχο αυτό. Ε, το κατά πόσον Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον ε, μπορούμε εμείς να αποσυρθούμε, αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι τα κράτη είναι αρκετά ισχυρά για να μπορέσουν ε, να σταθούν στα πόδια τους, αν θέλετε, μόνοι τους. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να, να αλλάξουμε άρδινε τα κράτα αυτά. Τώρα, από, από πλευράς περιφερειακής πολιτικής ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει μια δυναμική στην περιοχή αυτή που αποτελεί ένα, μια αντίχηση, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τουλάχιστον σε μακροοικονομικό επίπεδο. Έτσι το είδα και εγώ όταν ξεκίνησα την έκθεση αυτή. Όντως υπάρχει μία μίμηση, αν θέλετε, ή μία ε, ε, μια επίδραση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική της περιοχής και των κρατών. Τώρα βέβαια πιστεύω ότι όλα όσα προσπαθούμε να κάνουμε δεν μπορούν να γίνουν ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι από τη μία μέρα στην άλλη η περιοχή της, του Σαχέλ θα γίνει μια περιοχή ανθυρή που θα μπορέσει να συνδιαλλαγεί επίσης όρις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε και τι έχουν γίνει και με τι, ποιο είναι το αποτέλεσμα και των συμφωνιών ε, του Κοτονού. Να δούμε πώς ε, προχωρούν και τα προγράμματα δράσης του Σαχέλ για τις χώρες Σαχέλ τις ίδιες. Και θα πρέπει να δούμε και το πρόγραμμα δράσης του ENP Τώρα, για τη δεύτερη ερώτηση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όσον αφορά την ε, ανάγκη να ενδυναμώσουμε την δημοκρατική εκπαίδευση και την δημοκρατική κουλτούρα στην περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την αδυναμία πολλών κρατικών υποδομών στο Μαλί κυρίως, όπου υπάρχει η χειρότερη ε, κατάσταση όσον αφορά την φιλητική ε, ισότητα, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι γυναίκες να εκπαιδεύονται, να καταρτίζονται κτλ. Τώρα, αν θέλετε να έχουμε ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πρόγραμμα δράσης ε, για κάθε περιοχή του Σαχέλ, πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση και πρακτική, δηλαδή παραδείγματο χάρη καλλιέργεια, γεωργικές καλλιέργειες ή και ε, ε, εκπαίδευση στα θέματα δημοκρατίας. Θα ήθελα να απαντήσω στην τέταρτη ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση δεν με αφορά για το γραφείο της Δυτικής ε, Αφρικής. Όντως το πραξικόπημα στο Μαλί ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να είχε συμβεί. και καλό ήταν που έχουν γίνει οι εκλογές, που ε, οργανώνονται εκλογές και οργανώθηκαν εκλογές για την αλλαγή της κυβέρνησης. Το λόγο τον έχει ο Αλεξάνδρ. Ευτό για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και σχόλια. Θα μιλήσω πολύ ε, ε, η απάντησή μου θα στηρίζεται στα θέματα πολιτικής ορθότητας ή το ανάποδο. Το θέμα ποιο είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε σαφείς για τα δημογραφικά θέματα και αν θέλεις να περιορίσεις τη δημογραφική πίεση, τότε έχεις μεγάλη πιθανότητα να προσβάλλεις, να θίξεις κάποιον. Και επειδή δεν είμαστε και ειδικοί στα δημογραφικά θέματα, δεν έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά που κάνουμε. Έχετε απόλυτα δίκιο όμως όταν λέτε ότι αν το δημογραφικό προφίλ μιας χώρας διπλασιάζεται κάθε δεκαετία, τότε θα έχουμε όντως σοβαρό πρόβλημα, διότι όσο και αναπτυγεί ό,τι αναπτυξιακή βοήθεια δίδεται ε, θα πάει στράφη. Μην ανησυχείτε, λέει ο κύριος Γκέρενς, ε, ε, το ίδιο σημαίνει και στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, να σας πω να σας παρουσιάσω κάποιες, ε, κάποια στοιχεία δυναμικής ε, από, την, ε, από το Μαλί. Η Γαλλία πριν από δύο χρόνια είχε πει ότι έπρεπε να πάνε στρατηγικοί ακόλουθοι και σύμβουλοι για να βοηθήσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις του Μαλί να ενισχύσουν τις βόρειες περιοχές, τις βόρειες επαρχίες οι οποίες δεν μπορούσαν να, δεν μπορούσαν να τις διοικήσουν. Ήταν ακυβέρνητες. Και εμεί είπαμε ότι αυτό δεν, δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Ούτε στρατιωτική βοήθεια υπήρχε για το Μαλί και οι στρατιωτικές ε, δυνάμεις ε, του Μαλί πήγανε μόνες τους στην, ε, στις βόρειες περιοχές σε μια αδύνατη αποστολή, αν θέλετε μια αποστολή καταδικασμένη να αποτύχει και όντως οι απώλειες ήταν τεράστιες. Όταν υπάρχει, υπάρχουν τεράστιες απώλειες στο στρατό, αυτό δεν είναι καλό για το ηθικό του στρατού. Και ακολούθησε το πραξικόπημα. Το πρόβλημα τι, που, ήταν, που έχουμε τώρα είναι τι έπρεπε να κάνουμε. Ε, όλα να γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα έπρεπε να υπάρχει μια κατανομή αρμοδιότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη Τώρα συζητάμε το, τον πυρήνα του, το προβλήματος, χάρη το ρόλο ο, της, της Αλγερίας ε, μέσα στα πλαίσια της κοινή ε, ευρωπαϊκής πολιτικής α, ε, άμυνας και ασφάλειας, αλλά πρέπει να πούμε ότι τα χάλια στα οποία αντιμετωπίζει η περιοχή οφείλονται στην παρέμβασή μας στην περιοχή στη Λιβύη, διότι όλοι αυτοί του να είναι άνεργοι όταν εμείς εξαφανίσαμε τον εργοδότη τους, τον Καντάφη. Και η Γαλλία είπε σαφέστατα ότι έχουμε ένα μείζον ενδιαφέρον στην περιοχή, γιατί υπάρχει το ουράνιο. Αλλά δεν είναι μόνο οι Γάλλοι που έχουν ενδιαφέροντα στην περιοχή και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί ε, είχαμε απαγωγές ε, στην περιοχή από πολίτες αυτών των χωρών. Επομένως, είναι και ένα θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Προφανώς, εάν δεν συντονίσουμε την απάντησή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα υπάρχουν ε, δυσκολίες στον συγχρονισμό και στην ε, σύγκληση των διαφορετικών εθνικών ε, πολιτικών. Αλλά και ίσως τώρα να είναι λίγο καθυστερημένη η ζήτηση που γίνεται, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και ιδίω του συγγραφείς αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας έκθεσης. Δυστυχώς ο χρόνος θα αναγκάζει να ολοκληρώσουμε εδώ, αλλά πριν το κάνω αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή υπενθύμηση, να σας υπενθυμίσω κάτι. Σήμερα, ε, όχι σήμερα, σχεδόν με αυτή την Τετάρτη, μεθαύριο, θα υπάρχει μια αντιπροσωπεία του Μαλή με δύο άτομα, εκ των οποίων τον κύριο, ε, ε, ο κύριος Αζαρίδη που είναι από την ε, κοινή αντιπροσωπεία και θα έρθει εδώ για να συζητήσουμε για τα θέματα ασφάλειας ε, για το Μαλί. Την Τετάρτη 5 με 6 θα γίνει η συζήτηση. Η γραμματεία θα σας το επιβεβαιώσει, αλλά θα ήθελα ταυτόχρονα και μετά από τη συζήτηση που είχαμε με το, για το ΣΑΧΕΛ να προσπαθήσετε να έρθετε σε αυτή τη συνάντηση, Τετάρτη 5 με 6, διότι πρόκειται για μια περιοχή που μας ενδιαφέρει άμεσα και ο κύριος Αζαρίντ θα έρθει την Τετάρτη μεθαύριο. Ωραία, θα επιβεβαιωθεί ξανά το σημείο αυτό. Και περνάμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στην... Ε, Κυρία Κέλλερ, η οποία ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας, που ήταν και αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολόκληρου, έτσι, στη 13η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, που έλαβε χώρα στο Κατάρ, στην Τόχα, 21 26 Απριλίου. Η αντιπροσωπεία της ΔΕΒΕ λοιπόν πήγε στην Τόχα και εκτός από την κυρία Κέλλερ ήταν και ο κύριος Ντόιζερ και ο κύριος ε, Γιάνναν Σαλόμ ε, των σοσιαλιστών δηλαδή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Κέλλερ για να μας τα παρουσιάσει όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντω ήμασταν τρεις από την ΔΕΒΕ στη διάσκεψη αυτή τη Ουγκτάντ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το 2008 στην Άκρα πήγε αντιπροσωπεία από την Επιτροπή μας ΙΝΤΑ. Αυτή τη φορά πήγε από την ΔΕΒΕ. Η ΟΚΤΑΤ, όπως ξέρετε, είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Οπότε φυσικά και η ΔΕΒΕ έχει θέση εκεί. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας γίνεται η διάσκεψη της UNCTAD που ονομάζεται Committee of the Whole μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια για να καθορίζει την ατζέντα της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Τι στόχους βάζει δηλαδή, τι σκοπεύει να κάνει κτλ. Το θέμα αυτή τη φορά ήταν ε, παγκοσμιοποίηση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προς μία οικονομική ε, ανάπτυξη αλλά και γενικότερη ανάπτυξη για όλους και βιώσιμη. Ήταν και η κυρία Κέοβα, η Επίτροπος, ήταν και ο κύριος Γκουστάβο Μαρτίν Πράντα που είναι Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ εκτός από τους τρεις της αντιπροσωπείας μας. Οργανώθηκαν διάφορα πάνελ όπου συμμετείχαμε για διάφορα επιμέρους θέματα. Εμείς συμμετείχαμε σε ένα που ήταν γυναίκες στην ανάπτυξη, υπήρχε και κοινό που παρακολουθούσε τις παρουσιάσεις μας. Υπήρξε και ζήτηση κοιλής τραπέζης για την ενίσχυση όλων των μορφών συνεργασίας για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Υπήρχε και ένα φόρουμ για την κοινωνία των πολιτών που οργάνωνε ένα σωρό έτσι, εκδηλώσεις. συμμετείχαμε και σε πολλά άλλα και σε δημοσιεύσεις κλπ. Και διμερώς υπήρξαν και επαφές με τον κύριο Ράντι για παράδειγμα που είναι πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής ε, Ένωσης. Πολλοί από εσά τον γνωρίζετε. Μιλήσαμε γενικά για την επιρροή των κοινοβουλίων, πώς τα κοινοβούλια επηρεάζουν τη δουλειά της UNCTAD, ποιος είναι ο δικός μας ρόλος στη διάσκεψη αυτή επίσης συζητήσαμε. Συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης. Εκεί συζητήσαμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν και συναντηθήκαμε και με τον Γενικό Γραμματέα της Ούγκταν που είναι ο κύριος Πανιτσπάκτη. Αυτό έγινε την Τρίτη. Και συναντηθήκαμε και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να υπάρξει αλληλοενημέρωση μεταξύ μας όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Δύο φορές συναντηθήκαμε και με τον κύριο Πράντα που είναι ο επικεφαλής ε, ε, προσωρινά της Αντιπροσωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μας ενημέρωσε με τα δικό μας αίτημα για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Το αποτέλεσμα τώρα που μας ενδιέφερε ήταν να δούμε τι θα πρόβλεπε η UNCTAD για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, τι θα συμπεριλάμβανε στο πρόγραμμά της. Τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, ήταν ένα θέμα. Υπήρξε μία ομάδα βιομηχανοποιημένων χωρών που θέλανε να βγει αυτό το θέμα, γιατί λέγανε ότι υπάρχουν άλλες υπηρεσίες στο ΕΕ και άλλα προγράμματα που ασχολούνται με αυτό. Η UNCTAD όμως είπε, και εγώ πιστεύω ότι σωστά, πως έχουν ειδική άποψη για τα θέματα της ε, χρηματοδότησης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και ο ρόλος των υπονάπτυξων παρέμεινε. Εμείς πάντως, παρόλο που φάνηκε πως ε, αυτό θα ήταν καθοριστικό σε αυτήν την διάσκεψη, εμείς επιμείναμε ότι το θέμα της χρηματοδότησης έπρεπε να μείνει. Τελικά, οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν και η εντολή της UNCTAD παρέμεινε αρκετά ευρεία και ανοιχτή. Συνεπώς δεν ε, κόπηκε τίποτα από την εντολή ε, της UNCTAD και οι τρεις μας χαρήκαμε πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα ήταν καλό. Δόθηκε λοιπόν νέα εντολή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα δουλέψει βάσει αυτή τα επόμενα τέσσερα χρόνια UNCTAD. Τώρα δικός μας ο ρόλος ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ήταν κάπως περίεργο, γιατί συμμετείχαμε, όπως σας είπα, σε πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις και διασκέψεις, ακούσαμε ένα σωρό μιλητές, αλλά άλλο ρόλο δεν είχαμε. Μάθαμε πολλά. Πολύ ενδιαφέρουσες επαφές είχαμε. Δεν είχαμε όμως ένα ρόλο αυτό καθεαυτό, δηλαδή δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε ούτε την άποψη της Επιτροπής. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ίσως την επόμενη φορά, πριν την επόμενη διάσκεψη, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα πριν. Να δούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού κατευθύνεται, τι θέλει να πετύχει και να προσπαθήσουμε αυτό να το επηρεάσουμε πριν. Γιατί οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή και χώρες του Νότου ήρθαν και μας είπανε διάφορα για το ρόλο της Επιτροπής, δεν συμφωνούσαν. Άλλοι πάλι είπαν ότι έπαιζε ρόλο διαμεσολαβητή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι αλήθεια, καλό πάντως θα είναι την επόμενη φορά να ξέρουμε από πριν τι στόχους έχουν για να μπορούμε να τους επηρεάσουμε ανάλογα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στις επαφές με τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας ενημερώνουν για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας την προηγούμενη φορά είχαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ότι δεν είχαμε ενημερωθεί αρκετά. Αυτή τη φορά με τον κύριο Μάρτιν Πράτα συναντηθήκαμε δύο φορές. Ήταν πολύ θετικό, σίγουρα. Αλλά πάντα υπήρχε το πρόβλημα να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για την επόμενη επαφή, για την επόμενη ενημέρωσή μας. Και δεν υπήρξε συνέχεια μετά. Συνεπώς, παρόλο που είχαμε επίσημες επιστολές ε, από την Προεδρία, είχαμε επίσημη ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά υπήρξε πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την UNCTAD, έχει να κάνει γενικώ με τις διεθνείς διασκέψεις, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα άλλο ρόλο πέρα από το ρόλο του παρατηρητή. Να καθόμαστε εκεί, να παρατηρούμε τι γίνεται ε, και άντε λιγάκι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει, αλλά δεν συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις. Ίσως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά εφ' Υπήρχαν και άλλες αντιπροσωπείες του Φιλανδικού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα. Υπήρχε εκεί και ένας παρατηρητής από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή από την Νορβηγία υπήρχαν κοινοβουλευτικοί. Ίσως είναι πολύ καλύτερο αν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός με την κοινωνία των πολιτών. γιατί έτσι ίσως συμμετέχουμε καλύτερα, μια που δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην προετοιμασία, ούτε και στη συνέχεια που δίνεται μετά. Όπως σας είπα, μάθαμε πολλά για τα προβλήματα επίσης που έχει η UNCTAD, για τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την κοινοβουλευτική συμμετοχή και δίχως άλλο ήταν πολύ καρποφόρα η αντιπροσωπεία μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ και τους άλλους συμμετέχοντες, το προσωπικό που βοήθησε και που σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολο γι' αυτό να οργανώνει τις συναντήσεις μας εκεί. Μάθαμε πολλά, όπως σας είπα, και θα χρησιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ για την παρουσίασή σας αυτή. Δεν έχει ζητήσει κανένα το λόγο γι' αυτό και θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην SEAE, ε, ε, στην ε, Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Ευχαριστώ. Πίτερ Κρέμαν Πρέιτ. Είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας πριν έρθει ο κύριος Μαρτίν Πράντα επιτόπου ο μου. Θέλω και εγώ να σα δώσω τη δικιά μα εικόνα για τα αποτελέσματα τη διάσκεψης. Είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπό το φω των στόχων που είχαμε θέσει, στα συμπεράσματα τη προηγούμενη διάσκεψης, δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό βάσει και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Και αυτό που μας ε, απασχόλησε είναι η εντολή της UNCTAD να παραμείνει επικεντρωμένη, να μην είναι δηλαδή υπερβολικά ευρεία. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι η UNCTAD πρέπει να μείνει στην εντολή της, που είναι η ανάπτυξη και το εμπόριο και τα συναφή θέματα. Μας απασχολούσε δηλαδή αυτό να φανεί στο κείμενο. Αποσαφηνίστηκε στο κείμενο τελικά ότι η UNCTAD δουλεύει με τους πόρους που έχει στη διάθεσή της και σε συντονισμό με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Υπήρξαν θέματα που δεν θέλαμε να συμπεριληφθούν και συμπεριλήφθηκαν. Ήταν μια δύσκολη συζήτηση στο θέμα της πράσινης οικονομίας. Εμείς θέλαμε να γίνει μνήα στο ρόλο άλλων οργανώσεων, του IMF, του ILO, της Εθνούς Τράπεζας. Θέλαμε επίσης να υπάρξει μνήα της έλλειψης ποσοστώσεων και υπήρχαν και πολλές δυσκολίες για τα μονομερή μέτρα με την Κίνα, για παράδειγμα. Υπήρχαν πολλά θέματα που δεν θέλαμε να μπούμε στο κείμενο, όπως ήταν ο ρόλος της μεταφοράς τεχνολογίας, αντί για την έρευνα που θα στήριζε κάτι τέτοιο. Δεν θέλαμε να επεκταθεί η εντολή της Σούγκτατ σε δημοσιονομικά θέματα και δεν έγινε αυτό. Ούτε θέλαμε νέες οικονομικές υποχρεώσεις από τις ε, αναπτυγμένες χώρες μέσα στο κείμενο. Πιστεύουμε ότι το κείμενο είναι πιο συνεκτικό από ότι το προηγούμενο, στην προηγούμενη διάσκεψη και αυτό είναι θετικό. Πρέπει να υπάρχει ένα συνεχής όμως έλεγχος επίσης. Τελικά βρήκαμε μια λύση και τώρα ασχολούμαστε και κάνουμε διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, από τις οποίες είμαστε ικανοποιημένοι. Όσον αφορά τις σχέσεις τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακολουθούσαμε την ίδια προσέγγιση που ακολουθούμε και σε άλλες διεθνείς διασκέψεις. Σε συμφωνία με τη Συμφωνία Πλαίσιο δουλεύουμε και όπως και σε άλλες περιπτώσεις εμείς είμαστε στη διάθεση της αντιπροπίας του Κοινοβουλίου, ενημερώνουμε, δίνουμε στοιχεία. Είχαμε και δύο συναντήσεις με την αντιπροσωπεία σας, όπως είπε και η Ευρωβουλευτής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δίνουμε στοιχεία και πληροφορίες, όπως επίσης και για το πώς προχωράν οι διαπραγματεύσεις. Και όλα αυτά σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο που υπάρχει ανάμεσα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο που καθορίζει τους ρόλους μας εκατέρωθεν. Εμείς τηρήσαμε αυτή τη συμφωνία. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει και άλλα πράγματα, αλλά εμείς τηρήσαμε τη συμφωνία αυτή. Όσον αφορά την εκ των προτέρων ενημέρωση. υπήρχαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία ήταν στη διάθεση ολονών πριν από την διάσκεψη και βάσει αυτών των συμπερασμάτων δουλεύουμε κι εμείς. Άρα ήταν διαθέσιμα. όπως γίνεται και σε άλλες διασκέψεις στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα όπου η Κομισιόν μπορούσε να συναντηθεί εκ των προτέρων με την αντιπροσωπεία. Αυτή τη φορά η κυρία Γεωργίεβα ήθελε αλλά δεν ήταν εφικτό από πριν υπάρξει τέτοια συνάντηση της με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τόχα. Πρακτικά δεν γινότανε. Αλλά ο κύριος Μαρτίν Πράντα συναντήθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλερ, θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Εμείς την ερμηνεία ε, την συμφωνία πλαίσιο την βλέπουμε κάπως αλλιώς. Ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται ανα πάσα στιγμή. Αυτή είναι η δικιά μας ερμηνεία. Το ανα πάσα στιγμή για μας σημαίνει και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Αλλά όπως είπατε, εσείς τηρήσετε τις γενικές αρχές. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Σε κάθε διεθνή διάσκεψη πάντα έχουμε το ίδιο. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή γενικότερα. Και να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρχει συμφωνία από πλευράς και του Επιτρόπου του Αρμόδιου και του Συμβουλίου, γιατί την προηγούμενη φορά αυτή για το Συμβούλιο, να συμφωνήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, για παράδειγμα, εκ των προτέρων, για να ξέρουμε πότε θα συναντιόμαστε και ποιος θα κάνει τι. Σίγουρα και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα θα μπορούσε να ζητήσει από τον αρμόδιο επίτροπο πολύ πριν να έρχεται εδώ και να εξηγεί ποια γραμμή θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις. Ίσως και να εγκρίνουμε και κάποια ψηφίσματα εκ των προτέρων για να εξηγούμε ποια θα είναι η θέση μας ή ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι θα υποστηρίξει στις ε, συνεντεύξεις τύπου, για να μπορούμε κι εμείς να παρέμβουμε. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Ίσως δεν είναι εφικτό για όλες τις διεθνείς διασκέψεις, αλλά πρέπει να δούμε πού βάζουμε τις προτεραιότητές μας και εκεί να το φροντίσουμε. Η Επιτροπή από τη δικιά της την πλευρά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι κάπως πιο ανοιχτή και να ερμηνεύσει κάπως ευρύτερα αυτό που λέει η Συμφωνία Πλαίσιο, το at all times, ανα πάσα στιγμή. Αν έχετε μια θέση, θα πρέπει να προσπαθείτε να μας την περάσετε, να μας ενημερώσετε για αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κέλλερ για την απάντησή σας. Σύμφωνα επί της Εποφελούμε μάλιστα για να σας ευχαριστήσω για την δουλειά σας, την επιμονή σας, την παρουσία σας εδώ πάντα. Δυστυχώς για μας φεύγετε και πάτε στην Ίντα. Σίγουρα την οπτική γωνία της Επιτροπής ΔΕΒΕ δεν θα την χάσετε στην Ίντα που πάτε. Εκ μέρους όλων λοιπόν για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι μας λύβει το γεγονός ότι αποχωρείτε από την ΤΕΒΕ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία δεύτερη έκθεση επί αποστολής ε, του κυρίου Νιούτον ε, Ντάν ε, για την αποστολή στην Ινδία, δηλαδή λίγες μέρες μετά την συνάντηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ινδίας περιλάμβανε και τον κύριο Αρσένη, την κυρία Άστραμ και μένα προσωπικά και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Νιούτον Τζοντζ για να μας παρουσιάσει την έκθεση επί αυτής της αποστολής. Ε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που είσαστε εδώ διότι μπορείτε να με βοηθήσετε διότι από τους τέσσερις που ήταν στην Επιτροπή με την κυρία Σνίμπερ Τζάστραμ και τον κύριο Αρσένη δυο μας είμαστε εδώ σήμερα. Όντως πήγαμε στην ε, Ινδία 20 με 24 Φεβρουαρίου και ο, ο Επίτροπος Πίμπαλξ είχε ε, ζητήσει να υπάρξει μία αναθεώρηση της ενισχύσεως προς την Ινδία και υπάρχει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και ε, Ινδίας ε, που προχωράει και μπορεί να ολοκληρωθεί εφέτος. Άρα έχουμε πολλά να λέμε μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, αν δείτε κατά ε, την, έκθεσή μου καλύψαμε πολλά θέματα είχαμε πολλές συνεδριάσεις και σημαντικές και ενδιαφέρουσες και στο πρώτο ήμιση αναφέρομαι στις συναντήσεις με τους διαφόρους υπουργούς και δεν ξέρω αν κυρία Πρόεδρε διαφωνείτε μαζί μου αλλά ε, πιστεύω ότι οι συναντήσεις ε, αυτές ήταν ε, ναι μεν καλές οι οποίοι είπαν ότι αν θέλετε να μας ενισχύσετε στον ομοσπονδιακό πορυπολογισμό έχει καλός αλλά διαφορετικά εμείς είμαστε στην Ανιούσα και εσείς στην Κατιούσα στην Ευρώπη οπότε νομίζω ότι είχε δίκιο ο Επίτροπος Πίμπαλξ δεν υπάρχει λόγος να συμβάλλουμε στον τεράστιο προϋπολογισμό στο Νέο Δελχή διότι έχουν αρκετούς πόρους και δεν μας χρειάζονται στο επίπεδο αυτό αλλά συναντήσαμε και μη κυβερνητικές οργανώσεις πήγαμε σε διάφορα σημεία και ιδίω την Τετάρτη το πρωί είδαμε 60 εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών ήμασταν τέσσερις εκεί και αντιλαμβάνεστε ότι αφού είχαμε 60 άλλους συμμετέχοντες ε, έπρεπε να δουλέψουμε όλοι πολύ σκληρά και χαίρομαι που η γραμματεία ε, ε, πήρε καλά πρακτικά και ανέφερε τι συζητήθηκε. Μετά πήγαμε στο Ρατζαστάν, στην Έρημνο, σε διάφορα σημεία και είδαμε ότι εφόσον δεν θέλουμε να χρηματοδοτούμε τον ομοσπονδιακό προπολογισμό με την ευρωπαϊκή βοήθεια μπορούμε να βοηθήσουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους πανφτωχούς Ινδούς οι οποίοι ζουν μακριά από το Νέο Δελχή χωρίς ε, ηλεκτροδότηση, χωρίς τίποτα διότι μιλούσαμε ε, στο Σαχέλ για ένα εισόδημα ενός ευρώ την ημέρα και το ίδιο ο είναι και στην Ινδία. Οπότε ήδη έχουμε πολλές δυνατότητες να βοηθήσουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολλά προγράμματα και αυτά που είδαμε στο Ρατζαστάν στην ε, έρημο ε, ένα σταθμό υδροδότησης ήταν ε, πολύ χρήσιμος και χρησιμοποιήθηκε πολύ καλά. Ήταν λοιπόν μια εξαιρετική επίσκεψη. Είχαμε στο τέλος και ένα άλλο αξιοπερίεργο. Ο Κρήτον Αρσένης ερωτεύτηκε το κάρι, τρελαίνεται για κάρι, μπορεί να ρωτεύει και την Ινδία, αλλά εν πάση περιπτώσει για το φαγητό δοκίμασε όλες τις συνταγές κάρι και ελπίζω ότι αυτά είναι οι γενικές γραμμές για την ε, έκθεσή μας. Ε, ευχαριστώ, συμφωνώ, συναντήσατε πάρα πολύ κόσμο, συναντήσαμε ε, και μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός χρηματοδότηση ε, δεν ήταν εμπεκτικός αλλά ήταν στο μετέχνιο. Υπάρχουν βέβαια όλες οι κάστες στην Ινδία που ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες και εκεί όντως υπάρχουν δύο, αν όχι πολιτικές, κατηγορίες ατόμων. Έχουν μείνει δύο μόνο και πιστεύω ότι όσον αφορά την ανάπτυξη όντως δεν μας χρειάζονται πλέον αλλά για όλα αυτά τα άτομα δεν είναι όντως ανάπτυξη είναι κάτι μεταξύ ε, της ανθρωπιστικής βοηθείας και της αναπτύξεως αλλά δεν μας χρειάζονται πια στην Ινδία οι ηγέτες φροντίζουν οι διαφορές μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών να μην είναι τόσο οξίες αλλά δεν ε, το πράττουν, δεν μειώνουν το κενό και εγώ θεωρώ ότι ακόμη και αν η χώρα δεν μας χρειάζεται πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε μεγάλη φτώχεια χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς νερό ενώ υπάρχουν τα μέσα. Ο κύριος Γιάννης νομίζω ότι έχει κάποια ιδέα και θέλει να λάβει το λόγο. Χαίρομαι διότι αντιλαμβάνουμε ότι κάποιος ε, ε, προειδεάζεται για το τι επιθυμώ να κάνω. Έχω πει επανειλημμένως τι μπορούμε να κάνουμε στις χώρες που είναι υποανάπτυξη. Ε, ε, αυτές οι χώρες πρέπει να προβούν στη διαφοροποίηση που προβλέπεται εις ε, την ατζέντα της, του μέλλοντος Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μειώνουμε με τις προσδοκίες μας και κάπως απογοητεύομαι διότι αν θέλουμε όντως να πραγματοποιήσουμε τους στόχους θα πρέπει οι αναδιόμενες χώρες να μπορέσουν συγχρόνως να κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αλλάξουν την πολιτική τους να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει ένα, μια αλλαγή του παραδείγματος και σήμερα θα πρέπει να συνδυάσουμε με την εσωτερική αλληλεγγύη κάτι το οποίο μέχρι στιγμής ε, είχε επινοηθεί μόνο για εξωτερική αλληλεγγύη. Το επαναλαμβάνω κατά κόρον, αλλά το Σεπτέμβριο θα γίνει μια διάσκεψη για τους στόχους της ε, ε, χιλιετίας και θα ήθελα να ξέρω τι λένε οι αναδυόμενες χώρες επί του θέματος. Μπορούμε να συνδράμουμε, υπάρχουν ακόμη χώρες που δεν είναι αναδιόμενες και στην αρχή είχα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ε, οργάνωση μιας ειδική διασκέψεως επί του θέματος και θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια εκδήλωση για να υπενθυμίσουμε στον καθένα ποιες είναι οι ευθύνες του. Σύμφωνο γιατί αν μια χώρα αναδυόμενη δεν κάνει τίποτα εμείς τι θα κάνουμε όταν δεν μας θέλουν. Δεν μας θέλουν. Ε, σε εμά είναι η εσωτερική αλληλεγγύη η οποία επιδρά και στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και αλλού. Ε, θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιήσουμε άλλους πόρους οι οποίοι μπορούν να αντεπεξέλθουν αυτής της φτώχειας. Ας οργανώσουμε αυτή, αυτή τη διάσκεψη. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει η Κομισιόν εάν πρέπει να αναλάβει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά το έχουμε συζητήσει αρκετά νομίζω. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τώρα και στους άλλους ενδιαφερομένους, αλλά καλό θα είναι να συζητήσουμε για αυτή την διάσκεψη, γιατί και σε 10 χρόνια ε, τα ίδια, ίδια κατάσταση θα αντιμετωπίσουμε. Κοιτάξτε στην Ολομέλεια πέρασε μια σε μια ψηφοφορία ακριβώς αντίθετη με αυτό το οποίο λέω τώρα. Επομένως, εφόσον θέλει το Κοινοβούλιο να είναι συνεπές, ας αρχίσει να εφαρμόζει τη συνέπεια στον εαυτό του. Η κυρία Τέρινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς, μόλις, μόλις τώρα είδαμε την έκθεση, επομένως δεν μπορώ να απαντήσω και να σχολιάζω το περιεχόμενο της έκθεσης, επομένως επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες σκέψεις σε αυτά που ακούστηκαν στην αρχή. Η συνεργασία για ανάπτυξη που δίδει, αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε στην Ινδία και κάνουμε παραδοσιακά είναι τομεακά να ενισχύουμε ε, και δίνουμε αρκετά χρήματα. Παραδείγματο χάρη στον τομέα της εκπαίδευση έχουμε δώσει μισό εκατομμύριο ευρώ κατά διάρκεια κάποιων ετών, το ίδιο και για την υγεία. Πώς χρηματοδοτήθηκαν τα κονδύλια αυτά. Δώσαμε στην κυβέρνηση της Ινδίας ε, χρήματα μέσω των προγραμμάτων που ε, χρηματοδοτεί η ίδια η κυβέρνηση. Δηλαδή τα διαχειρίζεται κονδύλια αυτά η κυβέρνηση, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρή στον τρόπο που διαχειρίζεται τα κονδύλια αυτά και υπάρχει ένα στοιχείο ηχνηλασιμότητας αν θέλετε. Μπορεί ανα πάσα στιγμή να εντοπίσει πού βρίσκονται τα χρήματα και πού εδόθησαν. Και ήταν εύκολο να δούμε πού πήγαιναν τα χρήματα, πώς τα χρησιμοποίησαν Επίσης, αν λάβουμε υπόψη μας ε, τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας σε συνεργασία με άλλους χορηγούς ε, στην, στον τομέα αυτό, που είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, η Τράπεζα Ανάπτυξης, ε, βλέπετε δηλαδή ότι υπήρξε μια γενικότερη συνεργασία αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ξέρουμε που πάει τα χρήματα αυτά, έστω και αν έχουν δοθεί ανατομής και υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ε, και μέσω του ελεγκτικού μηχανισμού της κυβέρνησης της Ινδίας μπορούμε να παρακολουθήσουμε την διάθεση των κονδυλίων. Τώρα, ο επόμενος κύκλος ξεκινάει το 2014 δεν θα συνεχίσουμε ενδεχόμενα με αυτή την τομεακή ενίσχυση. Συμφωνούμε με τα βασικά επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν εδώ, ότι η Ινδία είναι μια αναδυόμενη οικονομία. Κανείς ε, δεν μπορεί βέβαια να αμφισβητήσει το γεγονός ότι υπάρχουν ε, Υπάρχουν, πάρα πολλοί φτωχοί στην Ινδία. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και τον ρόλο της Ινδίας σαν, ένας, σαν έναν παγκόσμιο παίκτη η Ινδία είναι μια, ένας αναπτυξιακός συνεργάτης ε, ο, η ίδια ε, και βοηθάει χώρες της περιοχής ε, της, Νεπάλα, Μπουτάν, Αφγανιστάν και ακολουθεί αν θέλετε και τον δρόμο της Κίνας και κοιτάει και την Αφρική. Επομένως η Ινδία γίνεται δωρητής η ίδια Επομένως, είναι λίγο περίεργο να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας συνεργασία στα μοντέλ, στο μοντέλο που ε, ίσχυε μέχρι τώρα. Ε, αν δείτε επίσης ε, και το στρατηγικό έγγραφο για την Ινδία, που κάλυπτε την, περιοχή, την περίοδο μας το 2014, λέμε σαφέστατα και με την, και με την υποστήριξη της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή η συνεργασία θα ολοκληρωθεί εδώ. Και λέμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε την προοπτική με την οποία να αντιμετωπίζουμε την Ινδία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και η Ινδία δεν θα εξασφαλίσει κάποια χρήματα από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποια κονδύλια, παραδείγματο χάρη, για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτές οι ΜΚΟ θα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Δημοκρατία ή για το περιβάλλον ενδεχόμενα και υπάρχουν ε, μη κυβερνικές που μπορούν να διεκδικήσουν τα κονδύλια αυτά. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο, αν θέλετε, που είναι το εργαλείο συνεργασίας και η Ινδία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα μπορεί να πάρει χρήματα από εκεί, αλλά αυτό θα ενισχύσει τη στρατηγική μας συνεργασία και θα, είναι, θα υπάρχει ένα στοιχείο αμοιβαίου συμφέροντος, αν θέλετε. Επίσης υπάρχει και η ανθρωπιστική βοήθεια που θα συνεχίσει εφόσον η Ινδία αντιμετωπίζει καταστροφές, όπως ε, έχει γίνει και στο παρελθόν. Η ΕΚΟ είναι ε, παρούσα και στο Τζαμού και Κασμίρ και σε πολιτείες γενικότερα που πλήττονται από κυκλώνες στο Ουταρ Πραντές. Είμαστε παρόντες και η Ινδία μπορεί να διεκδικήσει κάποια κονδύλια μέσα στα πλαίσια όμως της αμοιβαίας ενίσχυσης, εκεί, της διμερούς βοήθειας, εκεί θα πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν άλλες χώρες στην Ανατολική Ασία που χρειάζονται βοήθεια. Και νομίζω ότι είναι καλή είδηση το γεγονός ότι μπορούμε να στραφούμε τώρα και προς άλλες χώρες της περιοχής που είναι ακόμα φτωχές. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Νιούτον Ντάν. Να ευχαριστήσω πολύ για την απάντηση. Είναι καθυσικαστική. Ε, σκεφτόμαστε, είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο όσον αφορά κάποιες περιοχές. Δύο σύντομες ιστορίες μου ήρθαν στο μυαλό. Ίσως οι συνάδελφοι να θυμούνται ότι πριν από 18 μήνες είχε γίνει μεγάλη διαφήμιση για έναν Ινδό, ο οποίος ε, ξεκίνησε μια απεργία πείνας, διότι διαμαρτυρόταν κατά της ε, διαφθοράς ε, της κυβέρνησης των Δελχή, αλλά γενικότερα κατά της διαφθοράς. Και αποφάσισε να κάνει απεργία πείνης, πείνας και να πεθάνει εάν δεν σταμάταγε η διαφθορά στην Ινδία. Είχε πολλούς οπαδούς και πίστηκε να σταματήσει την ε, απεργία πείνας όταν η κυβέρνηση ε, του υποσχέθηκε ότι θα υποβάλει ένα νόμο κατά της διαφθοράς. Μάθαμε τώρα ότι και, τα δύο, και οι δύο βουλές και η Άνω και η Κάτω Βουλή της ε, Ινδίας απέρριψε το νομοσχέδιο αυτό. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι και πολύ δεσμευμένοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ινδία. Δεύτερον, Μήπως κάποιος θα μπορούσε να μας πει ποια είναι η πολιτική ανάπτυξη της Ινδίας, να μας δώσουν ένα κείμενο. Είσαστε μια αναδυόμενη υπερδύναμη όταν κάναμε αυτή την ερώτηση εμείς, ε, κανείς ε, δεν μπόρεσε να μας απαντήσει, το και ο κύριο Κραβίνιο που είναι ο πρέσβης μας εκεί, που μας βοήθησε τόσο πολύ. Δεν υπάρχει τέτοιο κείμενο. Έχω την αίσθηση επομένως ότι η βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια προς την Ινδία στρέφεται περισσότερο στην ασφάλειά της, έτσι ώστε αναφέρθηκαν διάφορες, ε, διάφορες ε, χώρες όπως ε, το Μπουτάν και τα λοιπά, εκεί οι παραμεθόριες χώρες, διότι η Ινδία ανησυχεί με το, για, με, για την Κίνα και για την πειρατεία στην, στον Ινδικό και ενισχύει τις ναυτικές της δυνάμεις. Και η Ινδία επίσης ανησυχεί για το Πακιστάν, για πολλούς και γνωστούς λόγους. Δεν υπάρχει όμως καμία βοήθεια τη Ινδία σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι περισσότερο πολιτική ασφάλειας έχει και όχι αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο στην παρουσίαση μιας μελέτης για την φιλοκτονία, έλλειψη γυναικών ή Πρόκειται για μια μελέτη που έχουμε ζητήσει μαζί με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Φιλοκτονία έχει μεταφραστεί το genericide στα γαλλικά και genericide στα αγγλικά. Φιλοκτονία λοιπόν. Πρόκειται για τη διάκριση σε βάρος των γυναικών. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε ως εξής. Είναι η τάση να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τις γυναίκες, να τους δίνουμε λιγότερη προσοχή, είτε πρόκειται για τη διατροφή τους, είτε πρόκειται για τις υπηρεσίες υγείας προς αυτές, είτε για την κοινωνική στήριξη. Και σε ορισμένε ε, χώρες αυτό οδηγεί στη μεγαλύτερη θρησιμότητα των γυναικών. Εκατομμύρια γυναίκες, είτε αυθόρμητα είτε υποεπίση, αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους για να επιλέγουν το φύλλο του παιδιού που θα κάνουν. Και έτσι να μην γεννάνε κορίτσια, γιατί τα κορίτσια θεωρούνται μερικές φορές βάρος για τις οικογένειες. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν έχει τις ρίζες του σε μια ε, πολιτιστική κουλτούρα ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων, κάτι το οποίο ενισχύει και το κλίμα βία σε βάρος των γυναικών με κοινωνικές συνέπειες, με δημογραφικές ανισορροπίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και που οδηγεί συχνά σε βία σε βάρος των γυναικών. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρίν Μπέζ πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν τη μελέτη μας για την φιλοκτονία. Συνδυάστηκε με ένα άλλο Ινστιτούτο του Ενωμένου Βασιλείου. Εγώ ονομάζομαι Κάρεν Μπίς και δουλεύω για ένα γερμανικό Ινστιτούτο. Πρώτα απ' όλα θα σας πω τα κύρια σημεία της παρουσίασής μου. Θα σας παρουσιάσω το φαινόμενο, θα σας δώσω και κάποιες ε, πληροφορίες και στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα θα σας πω τι συμβαίνει στην Κίνα, στην Ινδία και θα σας πω τι γίνεται και σε άλλες χώρες όπου υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Μετά θα σας δώσω τα συμπεράσματά μου και τις συστάσεις μου. Το 1990 Σεν έγραψε ότι πάνω από 100 εκατομμύρια γυναίκες λείπουν. Τι σημαίνει αυτό, ότι λείπουν. Για να το καταλάβετε αυτό, θέλω να σας δώσω κάποιους ορισμούς. Ο πιο σημαντικός είναι εκείνος της αναλογίας μεταξύ των δύο φίλων. Είναι οι άντρες προς τις γυναίκες και εκφράζεται είναι ο αριθμός ε, των αντρών για 100 για 1000 γυναίκες. Αυτό βέβαια μπορείτε να το δείτε σε διάφορους ε, ορισμούς. Μπορείτε να δείτε τι γίνεται στις γεννήσεις, πόσοι αγόρια γεννιούνται ανά 100 ή 1000 γυναίκες ή αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία. Επηρεάζεται βέβαια η αναλογία αυτή από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες μερικές φορές δεν ε, καταγράφονται ή σκοτώνονται μετά τη γέννα. Ή... Για διάφορους λόγους δεν μπορεί κανείς πολύ εύκολα να έχει ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Πολλές φορές πρόκειται για εκτιμήσεις μόνο. Τα ποσοστά που βλέπετε εδώ τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε κάθε χώρα του κόσμου όταν γεννιούνται τα παιδιά έχουμε περισσότερα αγόρια που γεννιούνται από ότι κορίτσια. Όμως σε χώρες όπου έχουμε την ίδια μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών, η θνησιμότητα των αγοριών είναι μεγαλύτερη από την θνησιμότητα των κοριτσιών. Για λόγους βιολογικούς λοιπόν φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ευάλωτες και κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν σε διάφορες ηλικίε. Τώρα, οι γυναίκες που λείπουν είναι η διαφορά ακριβώς ανάμεσα ε, στα δύο φύλλα σε διάφορες ηλικίε. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη της αναλογίας αυτής σε διάφορες χώρες. Οι χώρες που είναι μπλε είναι εκείνες όπου στη γέννηση έχετε 106 παραπάνω την αναλογία. Είναι οι χώρες δηλαδή όπου γεννιούνται περισσότερα αγόρια από ό,τι θα περιμέναμε κανονικά. Αν δείτε για το συνολικό πληθυσμό, βλέπετε και αυτό που σας είπα, ότι η σχέση αυτή εξισώνεται. Εξαρτάται βέβαια από την ηλικία του πληθυσμού, για να έχουν υπάρξει πόλεμοι ο συνολικός πληθυσμός είναι περισσότερο θηλυκού γένους παρά αρσενικού. Βλέπετε ότι υπάρχουν μερικές χώρες, το βλέπετε στο χάρτη αυτό, που η αναλογία αυτή είναι πάνω από 103. 103 αγόρια δηλαδή για 100 κορίτσια. Για διάφορους λόγους. Ο όρος της φιλοκτονίας χρησιμοποιήθηκε ε, αρχικά όταν πρόκειτο για θανάτωση ατόμων του ενός φίλου. Είναι πολύ δυνητός βέβαια. Θυμίζει τη γενοκτονία η φιλοκτονία. Όταν λέμε γενοκτονία, τι εννοούμε. Εννοούμε τις περιπτώσεις που ένα έθνος ε, σκοτώνεται επίτηδες. Στην περίπτωση της φιλοκτονίας είναι όταν υπάρχουν πρακτικές οι οποίες οδηγούν να επιλέγεται το ένα φύλλο σε βάρος του άλλου. Δηλαδή να προτιμάμε τα γόρια από τα κορίτσια. Κατά το παρελθόν αυτό γινόταν με πρακτικές ε, μετά τη γέννηση. Δηλαδή ότι ε, παραμελούσαμε τα κορίτσια. Τώρα όμως πρόκειται για μια πρακτική σε δύο στάδια. Πρώτα απ' όλα εντοπίζουμε το φύλλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά προχωράμε σε άμβλωση αν δεν θέλουμε το συγκεκριμένο φύλλο. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν πρόκειται για κορίτσι. Για ποιους λόγους γίνεται αυτή η επιλογή στο φύλλο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Δεν είναι μόνο ότι προτιμάνε οι τα αγόρια. Οι λόγοι είναι ιστορικοί και πολιτισμικοί. Έχει να κάνει σε πολλές χώρες και κοινωνίες με συνήθειες που είναι να θεωρούνται τα κορίτσια περισσότερο βάρος από ό,τι τα γόρια. Οικονομικοί λόγοι είναι μερικές φορές. Η κληρονομική Βλέπετε σε μερικές χώρες τα κορίτσια, οι γυναίκες, δεν μπορούν να κληρονομήσουν την περιουσία των γονιών τους. Οπότε οι γονείς βασίζονται στα γόρια. Ξέρουν ότι τα γόρια θα κληρονομήσουν την περιουσία τους. Οπότε τα προτιμάνε και τους δίνουν ό,τι οικονομική υποστήριξη μπορούν για να διασφαλίσουν και αυτή τα γερατιά τους μέσα από τα αγόρια τους. Οι γονείς Επίσης πρέπει να πρικοδοτούν τα κορίτσια, να παίρνουν πρίκα όταν παντρεύονται. Και αυτό είναι οικονομικό βάρος. Και αυτό είναι λοιπόν ένας άλλος ε, λόγος. Στην ε, Κίνα, στην Ινδία και αλλού οι πρακτικές αυτές αποφέρουν κέρδη σε όσους τις ε, θέτουν σε εφαρμογή. Υπάρχουν όπως είπαμε λοιπόν παραδόσεις, για παράδειγμα το όνομα περνάει στα αγόρια το όνομα των γονιών και όχι στα κορίτσια. Ένας άλλος λόγος που θέλω να αναφέρω είναι οι ισορροπίες στην οικογένεια. Έχει φανεί αυτό τα τελευταία χρόνια και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ότι οι οικογένειες έχουν την τάση να θέλουν μικρότερες οικογένειες. Αλλά να μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση της οικογένειάς τους. Αν έχουν ένα κορίτσι λοιπόν και θέλουν δεύτερο παιδί αλλά όχι παραπάνω, επιλέγουν να κάνουν αγόρι. Βέβαια στις διάφορες χώρες η κατάσταση είναι διαφορετική και όπως βλέπετε εδώ για παράδειγμα στο χάρτη η Κίνα και η Ινδία επηρεάζονται πάρα πολύ από το ζήτημα αυτό. Θα ξεκινήσω με την Ινδία. Στην Ινδία, κάτι που δείχνει το πρόβλημα αυτό, είναι όταν ε, κάνει κανείς κορίτσι και μεγαλώνει κορίτσι, είναι σαν να ποτίζει τον κήπο του γείτονά του. Αυτή είναι η παροιμία που ισχύει στην Ινδία. Στην Ινδία λοιπόν σήμερα υπάρχει μια αναλογία στη γέννηση 112 αγόρια κάθε 100 κορίτσια. Για κάθε 100 κορίτσια δηλαδή γεννιούνται 112 αγόρια μέχρι τα 15 είναι ακόμα μεγαλύτερο το νούμερο αυτό. Συνήθως μικραίνει, σε αυτή την περίπτωση όμως στην Ινδία αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο ευάλωτα τα κορίτσια στην Ινδία από ότι τα αγόρια. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η διαφορά. Αλλιώ θα έπρεπε να έχει μειωθεί αυτό το νούμερο. Και σε συνολικό πληθυσμό είναι 108 άντρες προς 100 γυναίκες. Η κατάσταση επίσης έχει επιδεινωθεί από το 1961 και μετά τότε έγινε κάποια απογραφή στην Ινδία. Στην Ινδία λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητα στις γυναίκες σε όλες τις ηλικίε, όχι μόνο για τα νεογέννητα ή πριν τη γέννηση. Σε όλες τις ηλικιακέ κατηγορίες έχουμε μεγάλη θνησιμότητα στις γυναίκες. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η διάκριση σε βάρος των γυναικών έχει καταργηθεί από το 61. Παρ' όλα αυτά, στις παραδόσεις πολλών οικογενειών έχει παραμείνει. Από το 1981, η αναλογία στην γέννηση έχει βελτιωθεί. Υπάρχει κάποια σταθεροποίηση. Στις μεγαλύτερες ηλικίες γυναικών έχει βελτιωθεί η αναλογία. Οι διακρίσεις γίνονται κυρίως πριν τη γέννηση. Αυτό που μας εκπλήσει επίσης όταν κοιτάμε τα στατιστικά στοιχεία είναι ότι η διάκριση του φύλου γίνεται κατά την εγκυμοσύνη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν μια οικογένεια έχει ήδη ένα κορίτσι ή όταν είναι να κάνει ένα πρώτο παιδί, τότε τα πράγματα είναι ισόρροπα. Αν όμως έχει ήδη ένα παιδί μια οικογένεια και το πρώτο παιδί είναι κορίτσι, τότε προσπαθεί για το δεύτερο να έχει αγόρι. Τον να υπάρχει όμως αυτή η ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων στα παιδιά μιας οικογένειας δεν είναι μια αρκετά καλή εξήγηση. Αυτό το οποίο επίσης μας εκπλήσει στην Ινδία είναι ότι οι πρακτικές αυτές επικεντρώνονται κυρίως στα νοικοκυριά, τα πιο εύπορα, με μεγαλύτερη εκπαίδευση. Θα περίμενε κανείς ότι δεν θα ήταν έτσι, όμως τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες συμμορφωμένες θέλουν μικρότερες οικογένειες, λιγότερα παιδιά δηλαδή, και άρα γίνονται αμβλώσεις για να αποφύγουν έναν επιθύμητο φίλο πιο συχνά. Επίσης επικεντρώνεται αυτή η διάκριση σε ορισμένες ε, περιοχές της Ινδίας. Μερικές φορές έχουμε 130 αγόρια για 100 κορίτσια που γεννιούνται ζώντα. Διαφέρει κατάσταση και ανάλογα με την θρησκεία. Η κατάσταση όσον αφορά τους ενήλικους βελτιώνεται. Η Ινδία έχει κάνει πολλά πράγματα για να βελτιώσει την κατάσταση. Και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό. Το 1994 υπήρξε η... ο προγεννητικός έλεγχος υπάρχουν τέτοιε τεχνικέ οι οποίες όμως απαγορεύουν την επιλογή του φίλου. Δηλαδή με, αυτές, με αυτό το προγενετικό έλεγχο δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει το φίλο του παιδιού πριν τη γέννηση. Απαγορεύεται. Τέτοια μηχανήματα δεν δίνονται παρά μόνο σε όσους έχουν συμφωνήσει με αυτούς τους κανόνες. Ο αντίκτυπος είναι θετικός. Γι' αυτό και ίσως παραμένει σταθερή κατάσταση, αλλιώς θα έχει επιδεινωθεί σε βάρος των γυναικών. Επίσης δίνονται οικονομικά κίνητρα για την μόρφωση των ε, κοριτσιών στις πιο φτωχές οικογένειες. Όπως επίσης υπάρχουν και προγράμματα για τους ηλικιωμένους. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν κάποιες επιπτώσεις, αλλά ο έλεγχος δεν είναι αρκετά καλός και είναι δύσκολο να πούμε σήμερα ότι μακροπρόθεσμα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τώρα θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την Κίνα. Και εδώ θα ξεκινήσω με μια παροιμία που δείχνει ποια είναι η κατάσταση στην Κίνα, ότι μοιάζει με αυτή στην Ινδία. Τα κορίτσια πάλι είναι σαν νερό το οποίο φεύγει από την οικογένεια και που δεν μπορεί κανείς να πάρει πίσω μετά το γάμο. Εδώ η αναλογία είναι 113 αγόρια για 100 κορίτσια που γεννιούνται. Δηλαδή είναι πιο έντονο το πρόβλημα εδώ. Στις ηλικίες κάτω των 15 είναι 117 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια στον πληθυσμό. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κορίτσια πεθαίνουν πιο συχνά σε νερή ηλικία από ότι τα αγόρια. Επίσης η επιλογή του φίλου είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στις παραδόσεις της κοινωνίας εκεί. Είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα παρόν και σήμερα. Ένα μεγάλο λόγο βέβαια για τη διάκριση αυτή σε βάρο των κοριτσιών είναι η πολιτική τη ε, Κίνα από το 1979 που ήταν η πολιτική του ενό παιδιού ανεκογένεια. Και ίσχυε το 60% του πληθυσμού στην Κίνα. Οι υπολογισμοί έχουν δείξει ότι η πολιτική αυτή είναι υπεύθυνη για το 50% όλων των κοριτσιών που, όπως λέμε, λείπουν από την κινέζικη κοινωνία. Λείπουν εντός εισαγωγικών. Αυτό που διαφέρει σε σχέση με την Ινδία είναι ότι στην Κίνα η αναλογία αυτή οφείλεται σε προγεννητικούς ε, παράγοντες. Στην Κίνα δεν είναι τόσο δηλαδή μεγάλες ηλικίε, είναι κυρίως πριν την γέννα που γίνεται η διάκριση αυτή. Κατά τα άλλα, όπως και στην ε, Ινδία, βλέπουμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο πρώτο παιδί και το δεύτερο παιδί. Στο πρώτο παιδί η αναλογία δεν διαφέρει ιδιαίτερα, ενώ για το δεύτερο παιδί διαφέρει πολύ. Στην Κίνα 41 εκατομμύρια κορίτσια λείπουν Η συνέπεια βέβαια είναι η κακή μεταχείριση των κοριτσιών, αλλά θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Και η Κίνα πήρε μέτρα για να αλλάξει η κατάσταση, γιατί η χώρα το βλέπει το πρόβλημα. Το 1995 υπήρξε μια νομοθεσία για, την, για τις αυλώσεις που γίνονται εξαιτία του φύλου και υπήρξε μια εκστρατεία «Μοιαζόμαστε για τα κορίτσια» υπέρ μια πολιτικής δηλαδή υπέρ δύο κοριτσιών εν οικογένεια, υπέρ της μόρφωσης των κοριτσιών. Παρ' όλα αυτά, μικρέ ήταν οι επιπτώσεις. Το 2006 διαπιστώσαμε ότι γενικεύθηκε, ενώ στην αρχή ίσχυε μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιφέρειες. Care for Girls λοιπόν λεγόταν η εξτρετή αυτή και δεν ήταν η μόνη εκστρατεία υπέρ των κοριτσιών. Θα σας πω τώρα δύο λόγια για το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες εκτός Ινδίας και Κίνας. Με 100 από τα 100 εκατομμύρια που σας είπα πριν, τα 40 είναι στην Κίνα, αυτά που λείπουν δηλαδή, τα κορίτσια που λείπουν, αλλά το πρόβλημα αυτό πρέπει να ξέρετε ότι το έχουμε και στην Ευρώπη, το σε χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για παράδειγμα. Εδώ έχετε ένα κατάλογο ορισμένων χωρών, όπου γίνεται η επιλογή ανάλογα με το φύλλο. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει δηλαδή. Στη δεύτερη στήλη βλέπετε το 2012 στις γεννήσεις ποια ήταν η αναλογία η Αλβανία, η Ερμενία, η Ζερβετζάν και η Γεωργία. Βλέπετε ότι έχουν κατά τη γέννηση 111 ή και ακόμα παραπάνω αγόρια ανά 100 κορίτσια. Αυτό σημαίνει ότι και εκεί γίνονται αμβλώσεις εξαιτίας του φίλου του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί. Και στις χώρες αυτές, αν δείτε την αναλογία στις ηλικίες μέχρι τα 15, και εκεί βλέπετε ότι αυξάνει η αναλογία το ποσοστό αυτό. Και πάλι δηλαδή, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα σε νεαρή ηλικία από ότι τα αγόρια σε αυτές τις χώρες. Άλλα σημεία που υπάρχουν τέτοιες πρακτικές, η Ποσοχάρη Αφρική. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σε αυτές τις χώρες η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι στην Ινδία και την Κίνα, αλλά όχι πριν τη γέννηση, μετά την γέννηση. Στην Υποσαχάρια Αφρική φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ ψηλά επίπεδα θνησιμότητας των ε, κοριτσιών και των γυναικών σε όλες τις ηλικίε. Αυτό οφείλεται σε ασθένειες και σε διακρίσεις. Η ελονοσία, για παράδειγμα, πλήττει πιο πολύ τα κορίτσια. Οι υπηρεσίε υγεία που προσφέρονται στα κορίτσια είναι λιγότερε από ό,τι στα γόρια. Αλλά και το AIDS, βέβαια, που και αυτό θανατώνει ε, πάρα πολλές γυναίκες που είναι πιο ευάλωτες από ότι οι άντρες αυτό. Κάτι ενδιαφέρον αλλά και απειλητικό συγχρόνως είναι ότι αυτέ αυτές οι ανισορροπίες που καταγράφονται στην Ινδία και την Κίνα είναι παρούσες και σε κάποιες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά ακόμα. Σε μερικές κατηγορίες δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχες αναλογίες όπως και στην Κίνα και στην Ινδία, μόνο που δεν αφορούν τον γενικό πληθυσμό των χωρών αυτών, αλλά συγκεκριμένες ε, κατηγορίες. Η Κορέα είναι μια, η Νότια Κορέα είναι μια άλλη περίπτωση η οποία είχε τέτοια φαινόμενα, πήρε δράσεις, απαγόρευσε τις αμβλώσεις εξαιτίας του φύλου και έκανε πάρα πολλές εκστρατείες και φρόντισε να στηρίξει τις οικογένειες με κορίτσια. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από το 2011 η αναλογία είναι περίπου φυσιολογική. Πέρσι επιτρέπηκε και πάλι να μπορούν οι γορείς να γνωρίζουν το φύλλο του παιδιού τους που θα γεννηθεί πριν τη γέννησή του, που σημαίνει ότι έχουν εμπιστοσύνη οι αρχές ότι οι οικογένειες δεν θα προχωρήσουν ε, σε τέτοιες φιλοκτονικές πρακτικές. Ποιες είναι οι συνέπειες? Κάποιες τις ανέφερα και στην εισαγωγή μου. Περισσότεροι άντρες σε μια κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν ε, κοινωνικά προβλήματα για τους άντρες που φοβούνται ότι δεν θα βρουν σύζυγο ή μπορεί να οδηγήσουν και σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Σε χώρες που υπάρχει τέτοια αναλογία έχουν εντοπιστεί και βίες πρακτικές, μεγαλύτερη πορνεία ή ε, εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών αλλά και πιο έντονη παρουσία σεξουαλικά μεταδόσιμων ασθενειών. Υπάρχει μεγάλη πίεση στις γυναίκες, όπως καταλαβαίνετε, διότι στις πρακτικές αυτές καταλήγουν οι γυναίκες μετά από μεγάλη πίεση. Καμία γυναίκα από μόνη της δεν πάει και λέει ναι, ναι, εγώ θέλω να σκοτώσω το παιδί μου επειδή είναι κορίτσι. Η ψυχολογική πίεση λοιπόν είναι τεράστια και οδηγεί μερικές φορές και σε αυτοκτονίες σκεφτείτε και τα κορίτσια που γεννιούνται γνωρίζοντας ότι δεν είναι επιθυμητά. Ότι δεν τα θέλουν οι γονείς τους επειδή είναι κορίτσια. Καταλαβαίνετε η ψυχολογική πίεση υφίστανται αυτά. Οι οικογένειες μερικές φορές μπορεί να μην αποφύγουν τη γέννηση ενός κοριτσιού, αλλά να το κρύβουν, να αποφεύγουν να το δείξουν για παράδειγμα, για να μην τις κατηγορήσει κανείς. Θα τελειώσω με κάποια συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις γενικά πρώτα και μετά συγκεκριμένα για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι μπορεί να κάνει. Είδαμε λοιπόν ότι στην Κίνα και στην Ινδία η αναλογία αυτή αυξάνει. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση αργότερα, αλλά σίγουρα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία βελτίωσης της κατάστασης. Δύο πράγματα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το ένα είναι η νομοθεσία και το άλλο είναι να αντιμετωπιστούν οι πηγές, οι αιτίες που οδηγούν στην επιλογή του φίλου του παιδιού. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό σε ολόκληρη την Ινδία ή σε ολόκληρη την Κίνα, σε ορισμένες περιοχές. Δύσκολα βέβαια μπορούμε να συγκεντρώσουμε αξιόπιστα στοιχεία. Μπορούμε να μετρήσουμε τα κορίτσια που γεννιούνται, αλλά όχι αυτά που δεν γεννιούνται για παράδειγμα. Μπορεί να μην ξέρουμε όλες τις ε, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για αυτές. Πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο και το θέμα των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν στην ε, στο φαινόμενο αυτό της φιλοκτονίας. Πρέπει επίσης να δούμε και τις συνέπειες στην υγεία, τις κοινωνικές, του φαινομένου δηλαδή που μας οδηγεί να έχουμε περισσότερα γόρια από κορίτσια, περισσότερους άντρες από γυναίκες και τι πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν που θα στηρίξουν την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Χρειάζεται επίσης να εκπονηθεί παρετέρω νομοθεσίες που να προβλέπει μεγαλύτερες κυρώσεις οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται δεν δίθεται πάντα σε εφαρμογή. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη ενημέρωση και πιο πολύ lobbying, πίεση προς τους γιατρούς, οι οποίοι υποφελούνται τελικά στις χώρες αυτές από την πρακτική. Κάποιε συστάσεις τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο από εδώ να επηρεάσει κανείς το τι γίνεται στην Ινδία και την Κίνα πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη για να αλλάξουμε τις πρακτικές αυτές που εφαρμόζονται στην Ασία. Θα συστήναμε οι επιτροπές σας να συνεργάζονται περισσότερο για να συμπεριλάβουν στα θέματά τους και στις συζητήσεις τους την έννοια αυτής των ε, αδύναμων γυναικών, των γυναικών που λείπουν από την κοινωνία μας. Έχει υπάρξει κοινή δήλωση από διάφορες, ε, διάφορους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών που μιλούν για αυτό το θέμα της επιλογής του φίλου Καλό θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη ή οι διάφορες, ε, διάφοροι οργανισμοί σε επίπεδο Ευρώπης να συνεργαστούν για να καταλήξουν σε κάτι αντίστοιχο. Επίσης να συμπεριλάβετε στα διάφορα προγράμματά σας με την ίδια την Κίνα να αναφέρετε πάντα την ανησυχία σας αυτή για το φαινόμενο. Όπως επίσης και σε κάθε μέσο αναπτυξιακό ή συνεργασίας Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για μεγαλύτερη συνδυτοποίηση του κόσμου και μέσα στην Ευρώπη και εκτός. Η Επιτροπή επίση για το Διεθνέ Εμπόριο θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν ρήτρε σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε που συνάπτονται με τρίτες χώρες ώστε να συμπεριλαμβάνουν αυτές και την ρήτρα αποφυγή του φαινομένου. Και να τονίζονται βέβαια και τα δικαιώματα των γυναικών. Τέλος, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει σε κάθε συνεργασία που έχουν να υπογραμμίζουν την ανησυχία τους για το φαινόμενο αυτό και να πιέζουν και διπλωματικά τις κυβερνήσεις των χωρών εκείνων που ανέχονται τέτοιες πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση και ξεκινώ με τον κύριο Μίτσελ ε, για τους παρεμβαίνοντες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την έκθεση γιατί ε, ήμουν εισηγητής για το θέμα αυτό και πράγματι εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν εμφανίζεται στην ετήσια έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο πριν μερικές εβδομάδες αλλά έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με τις διακρίσεις των φύλων που πρέπει να λύσουμε. Αν παίζαμε ε, ποδόσφαιρο μαζί θα βλέπαμε ότι έχουμε περισσότερα πράγματα που μας ενώνουν και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος στην Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις ε, από ό,τι νομίζουμε. Ε, σχετικά με τις διαφάνειές σας, τα παρουσιάσατε πολύ σωστά. Ελπίζω ότι θα είμαστε ενωμένοι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει το ένα κόμμα να εκμεταλλευτεί το θέμα έναντι ενός άλλου. Και το πρόβλημα είναι ότι λείπουν 100 ε, εκατομμύρια γυναίκες ε, στον κόσμο και στην ε, Ευρώπη πεθαίνουν 60 εκατομμύρια γυναίκες δεν είναι μόνο οι αμβλώσεις αλλά είναι και οι παιδοκτονίες και η εγκατάλειψη. Ε, είχαν υπάρξει σε μια εφημερίδα ορισμένα άρθρα επί του θέματος ε, όπου φαίνεται ότι όταν υπάρχει κορίτσι όλοι ενοχλούνται και είναι απαράδεκτο. Και έρχομαι σε ερωτήσεις μου τώρα κυρία Πρόεδρε. Νομίζουμε ότι αυτό συμβαίνει στις στοχές οικογένειες, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αποδείξατε στην έρευνα ότι στην ε, Ινδία συμβαίνει και στις εύπορες οικογένειες και τις πλέον ε, με μεγαλύτερη ε, παιδεία. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα στηρίξει τις προσπάθειές σας η Επιτροπή και εγώ θα ήθελα εδώ να πω Καταρχήν, μπορείτε να μας πείτε λίγο παραπάνω τι έκανε η Νότια Κορέα και πόσο εντατικά προσπάθησαν μέσω παιδείας, μέσω καταναγκασμού, δηλαδή τι δημιούργησαν, ποια ήταν η κίνηση που δημιούργησαν. Και νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο θέμα αυτό είναι ότι η οικονομική αξία ενός ε, άνδρα είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον θεωρείται μεγαλύτερη από τη μίας γυναίκας και από εκεί προέρχεται το παράδειγμα όπως και εσείς τονίσατε στη μελέτη σας. Άρα ένα θέμα που ίσως θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μετά το δεύτερο DCI είναι η ασφάλιση για τις καλλιέργειες γιατί αν καταστραφεί η καλλιέργειά σας ε, πρέπει να εξαρτάστε από τους γιους και ε, το θέμα της ασφάλισης γενικότερα και το συζήτησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Διότι πολλές φορές όταν μιλάμε για την Ασία, για τον υποανάπτυξη κόσμο, μιλάμε σαν να πρόκειται για κάποιον που είναι διαφορετικός από εμά. Και βλέπετε ότι στην Ασία τα παιδιά χειρίζονται καλύτερα τα κινητά τηλέφωνα από ό,τι εγώ ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν και ίσως ε, μπορεί να είμαστε εκτός θέματος λίγος, αλλά ε, νομίζω ότι η ασφάλεια είναι ουσιαστική. Η ασφάλεια ε, θα μπορούσε να βοηθήσει και να δούμε αν για οικονομικούς λόγους θα μπορούσε να βασιστεί κανείς περισσότερο στις νύφες από τις τους γιους και για την Κορέα ειδικά θα ήθελα να ξέρω ε, αν έχετε τα στοιχεία και μπορείτε να μου τα στείλετε τι είναι διότι είναι κάτι το οποίο στο Κοινοβούλιο πρέπει να μας απασχολήσει ε, στις επαφές με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τον ΟΗΕ, με το Συμβούλιο της Ευρώπης στα ε, στις ενώσεις ασιατικής φιλίας είναι θέματα που μπορούν να συζητούνται με κάθε ευκαιρία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ όντως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Με, με καταλαβαίνετε. Ανακαλύψαμε αριθμούς ε, οι οποίοι είναι τρομακτικοί. Και νομίζω ότι αυτή, αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός ενώ υπάρχει μια ε, συνθήκη για την αποφυγή κάθε διακρίσεως και υπάρχει διαφορά μεταξύ της αναγνώρισης ενός δικαιώματος και την εφαρμογή του. Θα ήθελα να πω εδώ ότι από το 1994 η διάκριση η οποία είχε παρουσιαστεί ε, και αυτή η πρακτική απαγορεύεται αλλά ε, το, την αντιμετωπίζουμε και στα κείμενα τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή δεν συνδυάζεται με κυρώσεις και δεν υπάρχει μία ε, δικαστική διαδικασία και άρα η κατάσταση είναι όντως απαράδεκτη. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς πέραν της Επιτροπής μας μπορούμε να φροντίσουμε το θέμα αυτό να συζητηθεί ε, πιο ευρέω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να προτείνουμε λύσεις, να προωθήσουμε τις λύσεις τις οποίες εσείς προτείνατε και άκουσα και με προσοχή αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μίτσελ. Δεν έχω άποψη σχετικά με την ασφάλιση, ίσως αξίζει να το ψάξουμε παραπάνω, αλλά είναι βέβαια ότι η οικονομική πτυχή είναι αποφασιστική σε αυτή την ε, ανισότητα. Και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιγκελ. Ευχαριστώ. Σήκωσα το χέρι μου την ώρα που νόμιζα ότι έχω κάτι να πω, το οποίο ίσως είναι διαφορετικό, όπως θα το πράξω τώρα. Γιατί άκουσα την έκθεσή σας ε, και αντελήφθηκα ότι παρουσιάζεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Συμφωνώ λοιπόν με την σύνοψή σας όπου υποδείξατε ορισμένα μέτρα, ορισμένες δραστηριότητες τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Ευρώπη. Και σήκωσα το χέρι μου διότι είμαι κάπως σκεπτικός για ορισμένα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε. Δηλαδή ήδη αισθανόμουν άσχημα διότι προφανώς συνέβαλα στη στατιστική σας. Εγώ έχω μόνο γιους, τρεις γιους. Αλλά διόρθωσα, απεκατέστησα τη βλάβη διότι οι γη μου έχουν έξι κόρες και κανένα γιο. και βλέπω ότι η χώρα μου, η Σλοβενία, είναι μία από τις αμφιλεγόμενες χώρες της στατιστικής σας. Αλλά δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω και η αντίδρασή μου είναι ότι ίσως έπρεπε να και λύσετε να μας βάλετε μπρος στον καθρέφτη και να μας πείτε ότι είμαστε εξίσου κακοί με τους άλλους, ίσως κάπως καλύτεροι, αλλά θα πρέπει να ε, ε, μοιραστούμε και εμείς την ευθύνη και να έχουμε το κρίμα στη συνείδησή μας. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν ευσταθούν οι υποψίες μου ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο κακή όπως ανέφεραν οι στατιστικές σας, διότι δεν μιλήσατε παραδείγματο χάρη, δεν ε, εστιαστήκατε συγκεκριμένα στις παραδόσεις και στις θρησκευτικές παραδόσεις και στην ε, θρησκεία ε, που παίζει ή όχι ε, κάποιο ρόλο στο θέμα και ευθύνεται η θρησκεία για αυτή την ανομαλία. Αν τώρα σκεφτώ την Ευρώπη και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν όμως πολύ σύντομα αυτά που μας είπατε δείξατε την ε, διαφάνεια και δεν ε, μπορούσα μετά να σκεφτώ που είναι οι επιφυλάξεις μου διότι ε, χωρίσατε στο το, τον κατάλογο ε, τη διαφάνεια σε διάφορα χρώματα. Εδώ βλέπω και τη Σλοβενία και έχω ορισμένα προβλήματα επ' αυτού και ίσως δεν εκφράστηκα σωστά. Θα χρειαζόμουν ε, περισσότερα επιχειρήματα διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί οι Ούγγροι δεν συμπαθούν τα κορίτσια ή οι Ιταλοί ή κάποιος. Εγώ δεν με πείθετε. Θα σας αφήσω να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε και άλλους τρεις ομιλητές και θα μαζευτούν πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με την τελευταία και μετά θα προχωρώ προς το πίσω. Σε αυτό το χάρη αυτός ο χάρτης δεν είναι τόσο καλός όσον αφορά τα χρώματα, γιατί μιλάμε για τις αναλογίες ε, ανάμεσα στα γόρια και στα κορίτσια. Ε, μπορεί οι περιοχές που έχουν κόκκινο να έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο, ας πούμε. Έχουν χαθεί πολλοί άντρες. Ε, ας πούμε, στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες, διότι πολλοί άντρες σκοτώθηκαν στον Δεύτερο Πόλεμο, ας πούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε περισσότερο, να δούμε περισσότερο με περισσότερες λεπτομέρειες. Πότε λείπουν γυναίκες, όταν γεννηθήκανε αργότερα, ε, πεθάνανε από ασθένεια, από αμέλεια, γιατί. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τη Σλοβενία, αλλά όπως και για την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και την Γεωργία, υπάρχει αυτή η διαφορά, αν θέλετε, διαφοροποίηση μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1991 είχαν ε, λογικές αναλογίες ανάμεσα στα γόρια και στα ε, κορίτσια. Μετά όμως σιγά σιγά άλλαξαν τα πράγματα. Μεταξύ αυτές οι χώρες μεταξύ τους έχουν και διαφορετικές ε, καταβολές, διαφορετική θρησκεία, πολιτιστικές πολιτιστικό παρελθόν και όχι δεν εμφανίστηκε όμως αυτό στι άλλες σοβιετικέ δημοκρατίες. Γι' αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε και να το ερευνήσουμε και να δούμε γιατί συνέβη. Επίσης υπάρχει και το θέμα της τρίτης γέννησης, του τρίτου παιδιού για ε, στην Ευρώπη, ας πούμε, για, τα, για το πρώτο και δεύτερο παιδί, οι αναλογίε είναι εντάξει, τα ποσοστά είναι σωστά. Μετά από το τρίτο παιδί και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Και δεν ξέρουμε να πούμε γιατί. Για τη δεύτερη ερώτητα, πόσο μπορεί να το συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα, μπορώ να σας πω ότι είναι καλό βήμα η σημερινή συζήτηση. Και όπως σας είπα, είναι σημαντικό οι διάφορες επιτροπές να συνεργάζονται. Και μπορεί να κάνουν την έρευνα και διάφορες επιτροπές. Δηλαδή, μία επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με κάποιους λόγους ή κάποιες πτυχές του προβλήματος και κάποιες συνέπειες του προβλήματος. Αλλά είναι σημαντικό κάποια επιτροπή να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην όλη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να το αναλάβετε αυτό, αν κάποιος θέλει να ηγηθεί αν θέλετε. Για την Κορέα τώρα να πω κάτι. It seems when you... Φαίνεται αν το δούμε έτσι γενικά, ότι στην Κορέα έχουν υιοθετήσει τα ίδια μέτρα όπως και στην Ινδία και στην Κίνα. Ένα πρόβλημα όμως είναι ότι η Κορέα έχει στην τελευταία 20 ετία μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Και σε μία μελέτη ε, ε, απεδείχθη ότι η προσωπική κατάσταση δεν αλλάζει την συμπεριφορά ε, του συνόλου. Δηλαδή, εάν μια οικογένεια γίνει πλούσια, δεν θα αλλάξει την συμπεριφορά της. Μονάχα εάν αλλάξει όλη η κοινωνία. Ας πούμε, στην Ινδία και πλούσια να είναι οικογένεια, δεν αλλάζει αντιμετώπιση. Στην Κορέα όμως, επειδή όλη η χώρα, όλη η κοινωνία πλούτησε, αναπτύχθηκε, τότε εκεί δεν στηρίζονται τόσο πολύ στα αγόρια. Και άλλαξε και η αντιμετώπιση τους απέναντι στα κορίτσια και στις γυναίκες εν γέννη. Πότε, πότε, πριν από 10 χρόνια, 20 χρόνια, ρώτησε ο κύριος Μίτσελ. Οι βελτιώσει εμφανίστηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια. Πριν από δέκα χρόνια η κατάσταση ήταν... Δεν έχω ακριβή νούμερα, ακριβούς, αριθμού, αριθμούς, αλλά πριν από 10 χρόνια ήταν όπως στην Κίνα και στην Ινδία. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει διαφορά στην Κορέα. Αλλάξαν τα πράγματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ναι, πολύ δύσκολο το θέμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον και περιμένουμε ανυπομονησία την έκθεση του κύριου Μίτσελ γιατί είναι περίπλοκο το πράγμα. Κάποιες σκέψεις μου, γιατί έχω πάει πολλές φορές στην Ινδία πρόσφατα, είναι όπως το σύστημα με τις κάστες. Η Ινδία, η Ινδία είναι ε, χωρισμένοι σε κάστες ε, κανονικά. Σου λένε όμως αν τους πεις κάτι για τις κάστες, α, εμείς έχουμε καταργήσει με νόμο το, τις κάστες. Αυτό όμως πρακτικά δεν έχει καταργηθεί. Στα χωριά ισχύει και, σε, και γενικά ισχύει. Θυμόσαστε κυρία Πρόεδρε, είμαστε μαζί στην Ινδία και συζητούσαμε με την Δήμαρχο για κάποια προβλήματα των τοπικών τοπικά και είχαμε μιλήσει για το θέμα ε, των ε, γυναικών που εξαφανίζονται και άκουσα μία γυναίκα ε, που είπε που είπε από πίσω μου, που έλεγε από πίσω μου έτσι ηρωνευτικά και κοροϊδευτικά, κανένα άντρα να αναλαμβάνει την ευθύνη εννοούσε να στραγγαλίσει το κοριτσάκι, το μωρό που μόλι γεννήθηκε. Τέλος πάντων, είχαμε πάει και σε μια περιοχή στο Μπιχάρ, όπου και εκεί συζητούσαμε ότι θα έπρεπε τα κορίτσια να μην παντρεύονται στα 13, γιατί επειδή είναι φτωχές οι οικογένειες εκεί, η μόνη δυνατότητα που έχουν για να ε, ε, επιβιώσει το κορίτσι είναι να το παντρέψουν νωρίς. Και, στην Ευρωπαϊκή, ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι αρκετά πετυχημένο, ε, εάν ένα παιδί, ένα κορίτσι δεν εγκαταλείψει το σχολείο στα 13 για να παντρευτεί και μείνει μέχρι τα 16, του δίνουμε ένα ποδήλατο. Είναι αρκετά πετυχημένο το πρόγραμμα. Τώρα, μια άλλη σκέψη μου. Επειδή έχω μια, μια μικρή γνώση της ιστορίας, πιστεύω ότι όταν μια χώρα έχει ένα πλεόνασμα ανδρών, τότε προχωράει σε πόλεμο. Και βλέπουμε τι γίνεται στην Ινδία και στην Κίνα. Έχουν πολύ περισσότερους άντρες από τι γυναίκες και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, μια και η Ινδία και η Κίνα ε, είναι αντίπαλοι και διεκδικούν τα νερά των Ιμαλαίων. Ε, και πιστεύω ότι αυτό εν δυνάμει μπορεί να είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω κύριε Μίτσερ αν πρέπει να το εξετάσετε και αυτό στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την... Uh, I will speak in Greek. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την, ε, το report που έχετε κάνει. Έχει πάρα πολύ σωστά στοιχεία μέσα. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω, κυρία Πρόεδρε, ότι η, από ιατρική απόψεως η σωστή αναλογία, η καταμετρημένη αναλογία είναι 106 αγόρια προ 100 κορίτσια και αυτό γιατί πράγματι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερο, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερου κινδύνου στην νεογνική ε, ηλικία και αυτό είναι καταμετρημένο σε όλε τι χώρε που έχουν σωστά στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει μια εξαίρεση, είναι η Αργεντινή, στην οποία έχει καταμετρηθεί ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεως γεννήσεων αγοριών. Αλλά και αυτό που έχουμε δει στην Ευρώπη, στις ε, Αζερβαϊτζάν, στην Γεωργία, στην, στα Βαλκάνια ίσως, ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ξεφεύγει προς το παθολογικό αν δεν, αν δεν μετρηθεί ταυτόχρονα και μείωση των γεννήσεων, μείωση του, ε, του πληθυσμού. Γι' αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα της Ευρώπης αυτό που περιγράφεται, αυτό που βλέπουμε 110 ε, αγόρια προς 100 κορίτσια. Το πρόβλημα είναι κυρίως στην Ινδία όπου το 2000 είχαν καταμετρηθεί 2 εκατομμύρια δολοφονίες νεογεννήτων, όχι εκτρώσεις, όχι αμβλώσεις. Μόλις είχαν γεννηθεί, είχαν, είχαν δολοφονηθεί 2 εκατομμύρια κοριτσάκια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που είπατε το sex selective abortion διότι όταν επιτρέπεται το abortion, όταν επιτρέπεται η άμβλωση, κανείς δεν θα πάει να ισχυριστεί ότι κάνει άμβλωση γιατί αφορά το φύλλο του παιδιού, καμιά δεν θα το κάνει αυτό. Συνεπώς είναι ζήτημα πια ρύθμιση των, των αμβλώσεων και όχι του sex selective abortion. Εκείνο που έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες είναι το sex selection αλλά μόνο στο επίπεδο του in vitro fertilization. Εκεί μπορεί να ισχύσει αυτό που μας έχετε πει. Τώρα, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο σωστό. Αυτό που κάνουν, σωστό, λάθος η έκφραση μου, αυτό που γίνεται σήμερα στην Ινδία είναι πιο κακό με τα ultrasound που προσδιορίζουν το φύλλο του παιδιού και κάνουν την άμβλωση στις πρώτες 6 εβδομάδες, 8 εβδομάδες ή να το αφήνουν να γεννιέται και να το δολοφονούν. Ή αυτό που γινόταν στην Κίνα με το ένα παιδί μόνο ήταν τόσο εγκληματικό σε σύγκριση με αυτό που γίνεται σήμερα. Άρα Εκείνο που πρέπει να γίνει και μας δώσατε πολύ σωστά το παράδειγμα της Κορέας είναι ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών αυτών αν θέλουμε να βελτιωθεί και αυτή η κατάσταση και όχι μόνο με ευχολόγια για την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά με ουσιαστικά μέτρα για την ε, για την λήψη όλων εκείνων των μέτρων, όλων εκείνων των παραγόντων που πραγματικά θα ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο. Γιατί σίγουρα και αυτό που είπατε ότι ένας άντρας δεν μπορεί να σκοτώσει ένα κοριτσάκι είναι και αυτό μέσα στην κουλτούρα που δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς από εδώ μέσα να διανοηθεί ότι υπάρχει το αντίδοτο ή το αντίβαρο σε οποιαδήποτε κρίση αξιών σε όλο τον κόσμο που θα επιτρέπει να κάνει κανείς αυτό το, αυτό το έγκλημα. Ευχαριστώ. Je vais terminer par Madame Bauer. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμάω όλος ιδιαίτερος την μελέτη και την έκθεση αυτή η οποία μας παρουσιάστηκε σήμερα. Και εκτιμώ όλους ιδιαίτερως την προφορική παρουσία που ακούσαμε. Η ερώτησή μου είναι εξή. Έχετε εξετάσει καθόλου τις αιτίε που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Υποθέτω ότι στην κάθε περιοχή στην οποία αναφέρεστε οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Δεν πρόκειται μόνο για την έλλειψη ασφάλειας. Σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες χώρες, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Οι γυναίκες δεν έχουν ε, δικαίωμα ιδιοκτησία στη γη. Οπότε οι οικογένειες, οι πλούσιες οικογένειες θέλουν να κρατήσουν την ιδιοκτησία και γι' αυτό προτιμούν να κάνουν αρσενικά παιδιά. Δεν ξέρω στην Ινδία τι ακριβώς ισχύει, Ξέρω όμως ότι σε άλλες χώρες της Ασίας, στην Κίνα για παράδειγμα, τα αρσενικά παιδιά, τα αγόρια είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν το μέλλον των γονιών, να βοηθήσουν δηλαδή τους γονείς όταν αυτοί φτάσουν στα γυρατιά τους. Έχετε λοιπόν πληροφορίες. Τι είναι αυτό που κάνει του, τους ανθρώπους να σκοτώνουν τα θηλυκά παιδιά, τα κορίτσια. Πιστεύω ότι είναι κάτι ευρύτερο. Είναι η κορυφή του παγόβονου αυτό το φαινόμενο, το, γενικό, το γεγονός δηλαδή ότι είτε σκοτώνονται τα κορίτσια είτε δεν τους προσφέρονται υπηρεσίες υγείας όπως προσφέρονται και στα αγόρια. Γνωρίζουμε τίποτα για όλα αυτά. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Έχουμε στοιχεία δεδομένα για την Κίνα και την Ινδία. Οι νόμοι δηλαδή που ισχύουν σε αυτές τις δύο χώρες στην πράξη πώς εφαρμόζονται. Όσοι καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές καταδικάζονται. Υπάρχουν νόμοι, αλλά οι νόμοι φαντάζομαι ότι δεν τηρούνται. Η εφαρμογή δηλαδή των νόμων δεν είναι καλή και έχω και μια παρατήρηση. Ο συνάδελφος Νιούτον Ντάν έκανε επίσης μια παρατήρηση και έχω ασχοληθεί και εγώ λιγάκι με την ε, εμπορία ανθρώπων. Η ιστορία μας δείχνει ότι στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μέχρι το 2020 και το 2030 μάλλον τον προηγούμενο αιώνα, είχαμε μεταφορά των γυναικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σιγά σιγά το εμπόριο αυτό γυναικών τη δεκαετία του 60 είχαμε ένα κύμα σαν για αυτό που έχουμε σήμερα ότι δηλαδή οι οικογένειες οι Πακιστανών για παράδειγμα στέλνουν τα κορίτσια τους 13-14 ετών σε οικογένειες προκειμένου να παντρευτούν στο τέλος. Είναι ένα σωρό περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε και θέλω να ρωτήσω αν όλα αυτά έχουν να κάνουν με την φιλοκτονία ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Όχι. Ποιος? Η Επιτροπή. Όχι. Κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Καλώς. Τότε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάλι θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Αναφέρθηκα πλήν στους οικονομικούς λόγους που οδηγούν στην επιλογή του φίλου μέσω της φιλοκτονίας. Σίγουρα τα κληρονομικά δικαιώματα αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως επίσης και η φροντίδα των ε, ηλικιωμένων. Η γυναίκα, το κορίτσι, άμα παντρευτεί, έχει υποχρέωση να βοηθάει τους γονείς του άντρα της. Για του δικού της τους γονείς πρέπει να το δεχτεί ο άντρα της για να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει κανείς που θα τους φροντίσει. Στην Νότια Κορέα αυτό που κάνανε ήταν ότι επέτρεψαν να υπάρχουν δικαιώματα των γυναικών ακόμα και μετά το γάμο. Δηλαδή μπορεί, έχει δικαίωμα η γυναίκα να φροντίσει τους γονείς της ακόμα και μετά το γάμο της. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, τα κληρονομικά δικαιώματα σίγουρα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά δεν ξέρω να σας πω ε, πού ακριβώς έχει υιοθετηθεί κάποιος νόμος κατά το φαινομένου αυτού ή όχι. Πάντως και στην Ιδία και στην Κίνα είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τέτοιες πρακτικές. Μια γυναίκα μπορεί να πάει σε ένα γιατρό και να δει ότι είναι έγκυος να μάθει το και μετά να πάει σε μια κλινική και να πει βιάστηκα. Οπότε θέλω άμβλωση, παρακαλώ. Συνεπώς. Τι άλλο, τι άλλο. Ορισμένοι νόμοι πράγματι δεν εφαρμόζονται καλά. Ένα πρόστιμο πληρώνει κανείς άμα παραβεί τον νόμο. Στην Κίνα πληρώνουν πρόστιμο για το δεύτερο παιδί, αλλά βλέπετε τι κάνουν. Θέλουν αγόρι. Οπότε προτιμούν, αν έχουν κάνει κορίτσι σαν πρώτο παιδί, προτιμούν να πληρώσουν το πρόστιμο, αλλά όντα σίγουροι ότι θα κάνουν αγόρι. Γιατί άμα είναι να κάνουν ένα δεύτερο κορίτσι, δεν θέλουν να πληρώσουν πρόστιμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η πολιτική της Κίνας που εξακολουθεί να ισχύει, που οδηγεί τελικά. Τώρα με τους... για τα στοιχεία, τα στατιστικά. Όντως, τα στοιχεία που έχουμε μερικές φορές ε, μπορεί να είναι ε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι γιατροί. Γιατί μερικές φορές δεν καταγράφουν τη γέννηση των κοριτσιών οι γιατροί, άρα τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε μπορεί να μην είναι απόλυτα αξιόπιστα. Παρ' όλα αυτά όμως, με τα στοιχεία που έχουμε τώρα, παρόλα αυτά σε χώρες όπως είναι το Αζερβαϊτζάν για παράδειγμα, για τα δύο πρώτα παιδιά υπάρχουν ε, κανονικές αναλογίες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Από το τρίτο παιδί και μετά αλλάζει η αναλογία αυτή. Άρα κάτι λένε τα νούμερα για την ύπαρξη διακρίσεων. Για την επιβίωση των βρεφών είναι ένα μεγάλο θέμα. Ε, ακόμα και όταν γεννηθεί ένα κορίτσι, ε, να ξέρετε ότι δεν παίρνουν την ίδια διατροφή τα κορίτσια και τα αγόρια. Ή άμα έχουν ένα παλτό, το δίνουν στα γόρια, όχι στο κορίτσι. Ή αν ένα κορίτσι είναι άρρωστο, δεν το πηγαίνω απαραίτητα στο γιατρό. Αν είναι ένα αγόρι άρρωστο, ναι. Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση δηλαδή και Εξού καταλήγουμε να μιλάμε για προτίμηση απέναντι στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Δεν είναι έτσι γενικά μου αρέσουν τα αγόρια και όχι τα κορίτσια. Οικονομικές στοιχείες. ναι, σας απάντησα για αυτές. Εντάξει, αυτά δεν έχω τίποτα άλλο. Ο κύριος Μίτσελ, κάτι ακόμα διάβασα πρόσφατα ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι το πρώτο παιδί είναι κορίτσι. Θέλει κανείς αγόρι όμως. Οπότε τι κάνει, κάνει δεύτερο παιδί. Και μετά όταν αποκτήσει πάλι κορίτσι, τι κάνει, δεν το θυλάζει ή δεν το ταΐζει καθόλου. Ενώ αν ήταν ε, αγόρι, θα το ταΐζει κανονικά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό ισχύει αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Χαίρομαι πάντως που μας φέρατε την έκθεση αυτή και φυσικά και πρέπει να συνεργαστούμε για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Λίγη συνεδρίαση αύριο το πρωί στην ίδια αίθουσα στις 9 για τους συντονιστές και στις 10 για τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλό βράδυ.